Um, their own proposals and uh, uh, uh, later initiatives. Dear Minister, thank you for coming. Um, it is a pleasure for us. And the floor is yours. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, κυρίες και κύριοι η σημερινή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να πω ότι είναι η τέταρτη επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που συμμετέχω τις τελευταίες δύο μέρες λόγω και του μεγάλου πορτφόλιου που έχω ως υπουργό. Ε, και συγκεκριμένα η παρουσία μου ενώπιον της Επιτροπής θα αποτελεί συνέχεια μιας... Συγγνώμη μας, ε, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Για τις προτεραιότητες και δράσεις που αναλαμβάνει να προωθήσει κατά τη διάρκεια τη εξάμεινη θητεία τη τα θέματα του διεθνέ εμπορίου. Όμω, πολύ πέραν τη ανταπόκριση μου σε καθιερωμένε πρακτικέ, η εδώ παρουσία μου είναι δηλωτική πράξη του σεβασμού απέναντι στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει για να διατηρήσει ή και να ισχυροποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα περισσότερο τη θέση τη στην παγκόσμια πολιτική σκηνή αλλά και για να καταστεί εσωτερικά μια δημοκρατικότερη οντότητα που αφουγκράζεται τους πολίτες. Άλλωστε κεντρικό μήνυμα και βασική προσπάθεια της Κυπριακής Προεδρίας είναι για μια καλύτερη Ευρώπη, πρώτα και κύρια για τους πολίτες της. Αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία λόγω της οικονομικής κρίσης. Ως απόρρια αυτής της κρίσης, Παρατηρούμε τους Ευρωπαίους πολίτες κάθε μέρα και πιο πολλοί να θέτουν υπό αφισβήτηση ακόμα και αυτό το οικοδόμημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το διεθνές εμπόριο, είτε όταν ασκείται στο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας, είτε σε διμερές επίπεδο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για αντιστροφή αυτής της κατάστασης, αφού αποτελεί ένα πυλώνα ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη και την αναθέρμανση της οικονομία. Θεωρούμε πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία ακριβώς συμβάλλουν ε, σε αυτήν την κατεύθυνση. Είναι παράλληλα όμως σαφές πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διατηρήσει την πρωτοπορία στην προάσπιση οικονομικών, οικουμενικών αρχών και αξιών, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, οι κανόνες δικαίου, η βιώσιμη ανάπτυξη και αυτές οι αρχές και αξίες να αντανακλούνται στις οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουμε σε διμερές επίπεδο, αλλά και στη συνεργασία μας σε πολυμερές επίπεδο. Αυτό άλλωστε αποτελεί υποχρέωση μας, η οποία πηγάζει και από το πλαίσιο στρατηγικής και το σχέδιο δράσης που πρόσφατα υιοθετήσαμε. Στην αρχική μου αυτή παρέμβαση συνοπτικά θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας πολιτικές και τα επιμέρους θέματα που θα διαχειριστούμε κατά τους επόμενους έξι μήνες, όπως συμφωνήθηκα στο πλαίσιο του τρίου, του τρίου της Προεδρίας. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την Πολωνική όσο και τη Δανική Προεδρία για τη συνεργασία που αναπτύξαμε όλη αυτή την περίοδο, αλλά και να τους συγχαρώ για την επιτυχή διαχείριση σημαντικών φακέλο που ανέλαβε. Ασφαλέστατα, η επίδευξη όλου αυτού του έργου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την επικοδομητική συνεργασία και σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, όπως επίσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αυτή σας τη συμβολή σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε. Ερχόμενο τώρα στα συγκεκριμένα θέματα. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συνεργασίας θεωρούμε πρόσφορο το έδαφος για επέκταση και εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων των χωρών της Νοτιού Μεσογείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν από την επιτάχυση των ε, εξελίξη διαπραγματεύσεων για τομεακές συμφωνίες, ευελπιστούμε στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών που βρίσκονται εξέλιξη, ώστε να ξεκινήσουν σύντομα διαπραγματεύσεις για σύναψη περιεκτικών συμφωνίων ελευθέρου εμπορίου με την Ορδανία, το Μαρόκο, και την Ισία. Όσον αφορά στι διμερεί συμφωνίε, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πω η περιεκτική οικονομική και εμπορική συμφωνία που επιδιώκουμε με τον Καναδά θα αποτελέσει μια από τι σημαντικότερε συμφωνίε που έχει συνάψει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν είναι η μεγαλύτερη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου παγκοσμίω. Η έκταση της, αλλά και οι πολλαπλοί τομεί που περιλαμβάνει, ανοίγουν πολλούς δρόμους για περαιτέρω οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη μεταξύ των δύο εταίρων. Δεν υποτιμούμε βέβαια τι εκκρεμότητε που παραμένουν σε σημαντικά θέματα και οι οποίε σχετίζονται με τι διαφορετικέ οικονομικέ δομέ και τα ρυθμιστικά συστήματα μεταξύ του Καναδά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, ευελπιστούμε ότι με καλή θέληση και διαλλακτικότητα οι εκτριμότητες αυτές θα επιληθούν εφόσον και οι δύο πλευρές εκφράζουν τη δέσμευσή τους για ολοκλήρωση της συμφωνίας. Σιγκαπούρη. Ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες της Ένωσης χωρών της Ασίας στην Ασία με την οποία έχω ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας ελευθέρων πορείου έχει επιδείξει την απαραίτητη θέληση και αφοσίωση για επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσει με τη Μαλαισία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ το Βιετνάμ, μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου, είναι η επόμενη χώρα Ασιαν, με την οποία έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσει. Αναφορικά με την ε, υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ινδία, η οποία λόγω του μεγέθους και του υψηλού ρυθμού ανάπτυξής της παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των υπηρεσιών, των επενδύσεων και των δημόσιων συμβάσεων. Από πλευρά μα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδο και να οδηγηθούν οι διαπραγματεύσει σε μια ισορροπημένη συμφωνία. Για να γίνει αυτό όμω είναι αναγκαίο να υπάρχει και η ανάλογη πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά, κάτι που μέχρι στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Δυστυχώ, οι διαπραγματεύσει με τι χώρε του Μέρκοσουα μετά την επανέναξή του αντιμετωπίζουν σημαντικέ προκλήσει, ιδιαίτερα μετά από τη σημαντική αύξηση από πλευρά Αργεντινή στη λήψη προστατευτικών προ τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει μέτρων, αλλά και λόγω και τη ε, στάση βεβαίω τη Αργεντινή ε, σε πολλά άλλα ζητήματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να δίνουμε τι προσπάθειε μα ώστε να παρηθούν αυτά τα μέτρα και οι διαπραγματεύσει να συνεχιστούν μέσα σε ένα επικοδομητικό κλίμα περαιτέρω μειώσεων των προστατευτικών ε, φραγμών. Επίση, στα πλαίσια τη ανατολική εταιρική σχέση, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τι διαπραγματεύσει για περιεκτικέ συμφωνέ ελευθέρων πορείου με την Αρμενία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, ευελπιστώντα σε ολοκλήρωσή του τον κατάλληλο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην υποβοήθηση της ανάπτυξης των απτυσσομένων χωρών επιδιώκοντας ένα διπλό αποτέλεσμα αφενός τη σταδιακή εσωμάτωση των χωρών αυτών στο παγκόσμιο εμπόριο και αφετέρου την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσα από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών ενδείκνυται η επιτάχυση των διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής χέρισης με τις χώρες της Αφρικής, Καραβακής και Ειρηνικού. Ω εκ τούτου, προσδοκούμε σε σταθερού ρυθμού πρόοδου για ολοκλήρωση συμφωνιών οικονομική εταιρική σχέση με περισσότερε από μια περιφέρεια των χωρών ΑΚΕ. Όπω γνωρίζετε, η διερευνητική μελέτη για μια συμφωνία ελευθερού εμπορίου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ιαπωνία έχει ολοκληρωθεί. Ο Επίτροπο Εμπορίου, κ. Δεκούχτ, στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου, έχει πληροφορήσει τα κράτη-μέλη ότι η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει σύντομα από το Συμβούλιο τη διαπραγματευτική εντολή για έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ακαλούθως το Συμβούλιο θα συζητήσει το θέμα και θα λάβει τις ανάλογες αποφάσεις. Ως Προεδρία θα διασφαλίσουμε ενεργώντας ως αξιόπιστοι διαμεσολαβητές ώστε το Συμβούλιο να καταλήξει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που θα αντανακλά το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμενοι τώρα στον σημαντικότερο εμπορικό μας εταίρο, τη ΣΥΠΑ, η προσπάθεια μας πρέπει να συνεχιστού, ώστε να διευκολύνουμε κάθε είδους συνεργασία που μπορεί να αποφέρει ωφέλη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η πρωτοβουλία σύστασης της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου με κύριο στόχο την εξέταση τρόπων ενίσχυσής της ε, της ενίσχυσής της, απασχόλησης και ανάπτυξης είναι ένα δείγμα. Θα έλεγα είναι δείγμα των δυνατοτήτων συνεργασία που υπάρχουν μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και που πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασία και ανάπτυξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένουμε τα αποτελέσματα τη μελέτη τη ομάδα εργασία και ανάλογα θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τι διαπραγματεύσει για τη σύναψη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τη ΣΥΠΑ. Όσον αφορά στην Κίνα, με την οποία οι εμπορικέ προοπτικές είναι σαφώ μεγάλε, διαφαίνεται ότι δημιουργείται σταδιακά το κατάλληλο κλίμα για ενδεχόμενη έναξη διαπραγματεύσεων για αυτόνομη επενδυτική συμφωνία. Φυσικά, όπω έχει αποδειχθεί διαχρονικά, η πολυμερή προσέγγιση των εμπορικών θεμάτων στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου μπορεί να δώσει άλλη διάσταση τόσο στι πολυμερέ εμπορικέ σχέσει όσο και στη δυναμική των διμερών σχέσεων. Για τον λόγο αυτό ευελπιστούμε στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εντός του τελευταίου εξαμήνου του έτους για αναζωγόνηση των διαπραγματεύσεων του γυρού της Δόχα εντός του 2013 με έφαση στη συμφωνία μέτρων υποβοηθητικών προς τις λιγότερα ανεπτυγμένες χώρε, στη διευκόλυνση του εμπορίου και στην αναθεώρηση των διατάξεων σχετικών με την επίλυση διαφορών. Πέραν των προαναφερόμενων, υπογραμμίζω το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα αριθμό νομοθετικών προτάσεων, όπως για παράδειγμα τις διμερείς ρήτρες διασφάλισης της Συμφωνίας της Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ε, Κεντρικής Αμερικής και στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Ε, θέλω σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι υπήρξε ε, η Κυπριακή Προεδρία προώθησε τα προσχέδια αποφάσεων του Συμβουλίου ε, και υπάρχει μια ομοφωνία σε αυτό το πράγμα, μια κατάληξη και αυτό είναι και ανταπόκριση βεβαίως στην επιστολή του Προέδρου της ΙΝΤΑ, ε, του Προφέσορ Μορέιρα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβαση που βοήθησε ώστε να επιταχυθούν τα πράγματα και ε, είναι θετικό το ότι σε αυτές τις λίγες μέρες η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να προχωρήσει αυτό το θέμα και να φτάσει σε μια έγκριση όπως βεβαίως ε, ε, οι προτάσεις της ε, Προεδρίας έχουν τύχει αυτής της έγκρισης και θα προωθηθούν. Επίσης, μπροστά μας είναι τα ζητήματα που αφορούν τις προτάσεις κανονισμών Omnibus 1 και Omnibus 2. Θέλω να πω ότι τέσσερα χρόνια μετά ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι αρκετά. Χρειάζεται να επισπεύσουμε αυτές τις διαδικασίες. Είναι ζητήματα που θα πρέπει ε, και είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα απασχολήσουν τους τριλόγους ε, για να προχωρήσουν και να προσπαθήσουμε ώστε να υπάρξει μια κατάληξη σε αυτές τις συμφωνίες. Στόχο στόχος μας δηλαδή είναι να επιτευχθεί συμφωνία για αυτούς τους κανονισμούς αν είναι δυνατόν πριν το τέλος του χρόνου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Πριν ε, δώσω το λόγο να σας πω πως ε, η Κυπριακή Προεδρία ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο πεδίο της εμπορικής πολιτικής πριν από λίγες ώρες ε, συνήθη συμφωνία στο πολύ ευαίσθητο επίμαχο θέμα το οποίο έχει τραβήξει πάρα πολύ δηλαδή τις εμπορικές προτιμήσεις ε, με το Πακιστάν. Βεβαίω είχε ήδη προχωρήσει πολύ το θέμα επί προεδρίας της Δανίας αλλά ξέρετε πως ε, πάρα πολύ συχνά το πιο δύσκολο είναι το να ε, κάνει κανείς τα τελευταία μέτρα. Και οφείλω να ευχαριστήσω την ε, Προεδρία της Κύπρου για το ότι κατάφερε να φτάσει σε έναν ισορροπημένο συμβασμό μαζί μας, σεβόμενη τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Δεύτερον και ίσως πιο σημαντικόν, η Προεδρία της Κύπρου μπόρεσε να πείσει το Συμβούλιο να συμβιβαστεί με το Κοινοβούλιο σε ένα άλλο επίμαχο και ευαίσθητο θέμα αυτό των εφαρμοστικών διατάξεων στα σχέδια συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την σύναψη εμπορικής συμφωνίας κάτι το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό καθώς το Κοινοβούλιο το ίδιο είχε καθυστερήσει να αντιδράσει και να καταλήξει σε μια κοινή θέση για το θέμα αυτό. Μπορώ να σας ανακοινώσω λοιπόν πως το Συμβούλιο σήμερα ενημέρωσε το Κοινοβούλιο πως ε, είναι διατεθειμένο να αφαιρέσει τις επίμαχες ε, πρόνοιες αυτές από τις ε, διατάξεις ε, του Συμβουλίου και να δούμε ακριβώς το πώς θα εφαρμοστούν οι συμφωνίες αυτές. Ε, αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο για μια προεδρία η οποία κάνει τα πρώτα της βήματα και νομίζω πως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τα επιτεύγματα αυτά. Αντιλαμβάνω πως το να έχει κανείς για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου είναι κάτι το πολύ απαιτητικό και συναρπαστικό. Γι' αυτό νομίζω πως ε, οφείλουμε να πούμε πως ε, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η Προεδρία και εύχομαι καλή επιτυχία και για την υπόλοιπη Προεδρία σας αλλά όσον αφορά την εμπορική πολιτική ήταν ε, εξαιρετική η αρχή που κάνετε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τώρα τη συζήτηση από τους ε, συντονιστές. Κάσπαρη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Έχω τρία θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ από ό,τι φαίνεται στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε για το μέσο πρόσβαση στην αγορά για την άσκηση πίεσης στις ε, χώρες ΑΚΕ και ανεξαρτήτως του εάν θα πάει το, στην Ολομέλεια τελικά το 2014-2015-2016 έχω την εντύπωση πως ε, καλό είναι να ασκήσουμε μια πίεση στους εμπορικούς μας εταίρους για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να μας βοηθήσει η Προεδρία του Συμβουλίου να ασκήσουμε και πίεση στην Κομισιόν, γιατί τα τελευταία χρόνια τις βλέπει αυτές τις διαπραγματεύσεις αποπέδει η Κομισιόν, οπότε πρέπει να ε, ασκήσουμε κάποια πίεση και βέβαια να επιδειχθεί και κάποια διάθεση συμβιβασμού. Οπότε θα θέλαμε τη στήριξη εδώ πέρα του Συμβουλίου. Κατόπιν αναφερθήκατε στις ε, διαπραγματεύσεις με το Mercosur. Ε, είναι διάφορο το ποιοι είναι οι λόγοι. Αυτό το οποίο κάνουν κάποιες κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή του Σούρ είναι περίεργο αν μιλήσουμε για την Αργεντινή ή τη Βραζιλία και θα ήθελα και να ενθαρρύνω πραγματικά την Προεδρία του Συμβουλίου και την Κομισιόν να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας στον ΠΟΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, γιατί νομίζω πως ε, Κανένας δεν μπορεί να λέει πως διαπραγματεύεται από τη μία συμφωνία εταιρική σχέσης και από την άλλη να ε, επιβάλλει καιρός οι οποίες δεν έχουν μία σχέση με το δίκαιο του ΠΟΕ. Και τρίτον, στον τομέα των διεθνών διαπραγματεύσεων, θίξατε το θέμα γενικά και από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή ε, τρέχουν γύρω στις 12 διαπραγματεύσεις ε, σύνδεσης, ε, ελευθερω εμπορίου κτλ. Και στις περισσότερες από αυτές δεν έχουμε διαπραγματεύσεις, έχουν κολλήσει κατ' ουσίαν. Και θα ήθελα εδώ πέρα η Προεδρία μαζί με Κοινοβούλιο και Κομισιόν να κάνει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων. Μιλήσατε για τις διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και προβλέπετε να ξεκινήσουν επόμενες διαπραγματεύσεις. Να σου πω δεν είναι δυνατόν να ε, ξεκινήσει 16ος, 17ος ε, ε, γύρος διαπραγματεύσεων για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τους Ιάπωνες για ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Εμείς ζητήσαμε να περιμένει το Συμβούλιο με την έκδοση διαπραγματευτικής εντολής μέχρι να εκφράσει την άποψή του το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να μας πει την άποψή σας γι' αυτό. Και το άλλο θέμα το οποίο αναφέρατε στον τομέα των Εθνών Συμφωνιών είναι η ΙΠΑ. Να σας το πω ξεκαθαρά, έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ πέρα. Αν δείτε το τι έχει κάνει και το Κοινοβούλιο στο παρελθόν, ήδη από το 2006 ζήτησε από την Κομισιόν από κοινού με τους Αμερικανούς να διαπραγματευτούν μια διατλαντική αγορά και να ολοκληρωθεί αυτή μέχρι το 2015. Δυστυχώς ε, έχουν περάσει έξι χρόνια, δεν έχει συμβεί σχεδόν τίποτα, έχουμε ακόμα τρία χρόνια μπροστά μας και θα ήθελα πραγματικά αυτό να αποτελέσει βασική προτεραιότητά σας η συμφωνία αυτή με τις ΗΠΑ. Νομίζω πως όλοι είδαν πώς ε, έχει εξελιχθεί η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 15-20 χρόνια, πόσο δραματικά μετατοπίστηκε το βάρος. Ε, ξαφνικά λοιπόν όταν μιλάμε για κανόνες, για προδιαγραφές, βλέπουμε πως οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην ε, Ασία, δοκιμάζουν τα όρια μας και θα πρέπει η ε, φιλελεύθερες δημοκρατίες πραγματικά να σχηματίσουν συμμαχίες και θέλω πραγματικά να δείτε αυτό το θέμα το διατλαντικό ως κορυφαία προτεραιότητά σας. Σας ευχαριστώ. Μπέντ Λάγκε, Σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Και εγώ θα ήθελα να σταθώ σε τρεις τομείς. πρώτα απ' όλα στο θέμα του πώς οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθοριστούν. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι η εμπορική πολιτική μας αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη, μόνο μέσα στο δικό της πλαίσιο και με τον τρόπο αυτό γίνονται συμφωνίες οι οποίες όμως οδηγούν να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Πριν από λίγες ώρες πήραμε μία απόφαση για το Πακιστάν στο Συμβούλιο, αλλά αυτό πρέπει να είναι και ένα παράδειγμα, ότι οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται με ένα τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχουν προβλήματα για θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Και εδώ υπήρξε ένα επιλεκτικό κατά κάποιο το πρόβλημα που αφορούσε μονάχα ορισμένε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά πιστεύω ότι οι θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να ενισχυθούν στην Ευρώπη μέσω της εμπορικής μας πολιτικής και αυτό θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο προτεραιότητας στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις που έχουμε και στις, πολυ... στις πολλές διαπραγματεύσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έρχομαι στο δεύτερο σημείο στην Ιαπωνία. Θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία με την Ιαπωνία, παραμένουν όμως σοβαρά ζητήματα κατά πόσο με τις τωρινές συνθήκες μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να επιτύχει τον στόχο της ενίσχυσης της απασχόλησης στην Ευρώπη. Και εδώ πάλι έχουμε το ερώτημα. Θα περιμένει το Συμβούλιο την άποψη του Κοινοβουλίου πριν δώσει τη διαπραγματευτική εντολή και θα θέσει την διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη ως ένα κεντρικό θέμα στη διαπραγματεύση με την Ιαπωνία. Τρίτος τομέας στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε στις ευκαιρίες που μας παρέχει η οικονομική μας σύνδεση με την Κίνα. Η δική μου εντύπωση το τελευταίο καιρό όμως είναι ότι η εμπορική πολιτική της Κίνας έχει περισσότερο σαν στόχο να προχωρήσει προς μια μεγαλύτερη, μια πιο ανταγωνιστική αν θέλετε σχέση με την Ευρώπη. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν πώς το Συμβούλιο θα μπορέσει μέσα στα, στο επόμενο εξάμεινο να ζητήσει από τους Κινέζους να έχουν μια πιο υπεύθυνη στάση. Παραδείγματο χάρη, μα σκεφτείτε τα θέματα των επιδοτήσεων τη Κίνα για, για τα φωτοβολταϊκά ή για τι αιωλικέ γεννήτριε, το γεγονό ότι παραγνωρίζουν και παραβιάζουν για πολλά προϊόντα τα πνευματικά δικαιώματα είναι σε πολλές περιπτώσεις ε, το μεγαλύτερο μέρος των παραποιημένων προϊόντων που έρχονται από την Κίνα ή τέλος και στα θέματα της πολιτικής πρώτων υλών που ακολουθεί η Κίνα. Πώς θα αντιμετωπίσει λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Ρόμπερτ Στέρντι από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι έχετε καλύψει ένα αριθμό συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου που έχουν έρθει στο προσκήνιο πρόσφατα και ανέφερε και ο Ντάνιελ ότι υπάρχουν και νέες τέτοιες συμφωνίες οι οποίες επίκυνται. Έχετε μία εξάμεινη προεδρία. Ποιες είναι οι συμφωνίες αυτού του είδους που θα θέλατε να τους δώσετε προτεραιότητα στο εξάμεινο της προεδρίας σας. Ποια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου απαιτεί την πιο μεγάλη προτεραιότητα από την πλευρά της Κυπριακής Προεδρίας. Δεύτερον, μία αποτελεσματική πολιτική εμπορίου δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς και κάποια μέτρα προάσπισης στον εμπορικό τομέα για να προστατευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ντάμπινγκ ή τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές άλλων χωρών. Ποιες είναι εδώ οι προτεραιότητες, τους, προτεραιότητες σας σε σχέση με τη διαδικασία εξυγχρονισμού των αμυντικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εμπόριο. Γιατί εγώ έχω εκπονήσει μια έκθεση πρωτοβουλίας ακριβώς για το θέμα αυτό. Ποιες είναι λοιπόν οι δικές σας προτεραιότητες για τα εμπορικά αντίμετρα που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα τώρα των Πρασίνων, ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο, η κυρία Κέλλερ. Αντικαθιστώ τον συντονιστή μας, δεν ξέρω αν ακολουθείτε μια σειρά ανάλογα με το μέγεθος των πολιτικών ομάδων. Αν και κανονικά οι πράσινοι είναι περισσότεροι από τους συντηρητικούς, απλά σας το τονίζω, όχι ότι έγινε και τίποτα όμως. Λοιπόν, έχω πολλές ερωτήσεις, θα περιοριστώ όμως λίγο, δεν έχουμε χρόνο. Για τον κύριο Υπουργό, θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία έχει καταλήξει το Συμβούλιο μετά από την ήττα την οποία ε, εν πάση περιπτώσει δέχτηκε στα πλαίσια της Συμφωνίας Άκτα και λόγω του περιεχομένου και λόγω της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε τι συμπεράσματα καταλήγεται για το Μερκοσούρ. Αναφερθήκατε ήδη. Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι λόγω της κατάστασης στην Παραγουάη η Παραγουάη αυτή τη στιγμή έχει εξαιρεθεί από τις διαπραγματεύσεις. Από την άλλη γνωρίζουμε ότι η Βενεζουέλα πρόσφατα έγινε πλήρες μέλος του Μερκοσούρ. Η χώρα αυτή τώρα θα συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις ή όχι. Και μια τελική ερώτηση. Η Κύπρος πράγματι βρίσκεται σε μια ειδική κατάσταση. Έχετε και εσωτερικό εμπόριο στα πλαίσια της πράσινης γραμμής, ανάμεσα στην Κυπρή Δημοκρατία, Κυπριακή Δημοκρατία και τον βορρά της νήσου. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα σε επίπεδο αυτό του εμπορίου για διάφορους λόγους, οι οποίοι δεν ακολουθούν πάντα μια κάποια λογική, αλλά έχετε πει ότι προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε τους πολίτες πριν από οτιδήποτε άλλο και γι' αυτό νομίζω ότι προς όφελος των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο Βορρά θα πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν από τις ρυθμίσεις αυτές. Θα πιέσει λοιπόν η Προεδρία σας για το άμεσο εμπόριο με τη Βόρεια Κύπρο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη δημοκρατία της Κύπρου. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό για τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Εντυπωσιακό ο κατάλογος των συμφωνιών και των ε, ρυθμίσεων στις οποίες αναφέρθηκε για το επόμενο εξάμεινο. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία συγκεκριμένα θέματα, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι. Θέματα που βρίσκω δύσκολα αλλά και ενδιαφέροντα. Πρώτον, για τον πολυμερή τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουμε στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτή την αντίληψη και θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε κάπως πιο συγκεκριμένα σχέδια έτσι ώστε να προχωρήσετε στα πλαίσια του γύρου DDA μέσα στον ΠΟΕ και στα πλαίσια των συμπερασμάτων της 7ης Υπουργικής Συνάντησης στη Γενέβη πέρυσι. Διαρωτώμε λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο Συμβούλιο θέλει να προωθήσει στα πλαίσια αυτά του ΠΟΕ. Και προφανώς αν γίνει κάτι τέτοιο το Κοινοβούλιο θα το ακολουθήσει με θετικό πνεύμα. Και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο θέμα που θα θέσω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συνομοθέτες. Διαρωτώ με εδώ. Το θέμα της εντολής για τις διαπραγματεύσεις είναι κάτι το οποίο σε μια πρώιμη φάση ε, θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους συνομοθέτες. Η εντολή βέβαια δίδεται από το Συμβούλιο, αλλά αν το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συνεισφέρει στον καθορισμό της κατεύθυνσης της εντολής των διαπραγματεύσεων των εμπορικών με τρίτες χώρες, τότε φοβάμαι ότι χάνονται και εμείς και εσείς το χρόνο σας. Γιατί όπως και στην περίπτωση της Άκτα, αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι το εμπόριο είναι προς όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίαρχα, ε, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί έτσι θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες ε, των πολιτών και του εκλογικού σώματος. Και ένα τρίτο θέμα τώρα. Αναφερθήκατε στις χώρες ΑΚΕ. Εγώ κατανοώ το πολυμερές εμπόριο σαν εικόνα της αναγνώρισης των αμοιβαίων συμφερόντων των εμπλεκομένων στην εμπορική αυτή συμφωνία. Εμείς είμαστε ένας από τους ε, εταίρους, από τους εμπλεκομένους. Πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια ατμόσφαιρα στο Συμβούλιο, έτσι ώστε να ανοιχτούμε καλύτερα για την αναδιοργάνωση των σχέσεών μας των εμπορικών στα πλαίσια των ΑΚΕ. Και ακόμα και με άλλες χώρες βέβαια, όπως η Ιαπωνία, η Ινδία και φυσικά οι χώρες Μερκοσούρ. Έχουν ζητήσει και άλλοι το λόγο. Η κυρία Μουσκαρντίνη. Ε, Παρακολούθησα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση την οποία έκανε ο κύριος υπουργό. Εγώ έχω την τύχη να, να πάω στην Κύπρο εδώ και λίγο καιρό και ξέρω και αναγνωρίζω την προσπάθεια με την οποία η κυβέρνηση της Κύπρου θέλει να ακούγεται η φωνή της στην Ευρώπη λόγω μια σειράς προβλημάτων που γνωρίζουμε καλά. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι πράγματι η ομάδα των Πρασίνων είναι μεγαλύτερη από, τους, ε, από την ομάδα των συντηρητικών και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζει καλύτερα την κατάσταση εκεί ε, πριν εκφραστεί στα θέματα τα εμπορικά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό της συγκεκριμένης χώρας και που οφείλονται σε δυσκολίες οι οποίες είναι γνωστές. Επανέρχομαι λοιπόν στα της ε, Κυπριακής Προεδρίας σε τρία συγκεκριμένα σημεία. Πράγματι δεν είναι πάρα πολλοί οι μήνες που έχετε μπροστά σας, ιδιαίτερα στο σημερινό πλαίσιο, το δύσκολο, στη σημερινή συγκυρία την δύσκολη, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για όλες τις γειτονικέ χώρες και λόγω ενός οικονομικού παγκοσμίου συστήματος το οποίο νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έχει χρονικά ε, εξοφλήσει θα έλεγα αυτό το καταναλωτικό ε, καπιταλιστικό μοντέλο το οποίο χρησιμοποιούμε έχει αποτύχει. Οι δυσκολίες λοιπόν είναι δεδομένες. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2010 το Κοινοβούλιο ψήφισε τον κανονισμό για τον καθορισμό προέλευσης των προϊόντων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, συνεισφορά και την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από αυτό το Συμβούλιο ε, δεν φαίνεται πουθενά. Ακούσαμε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που ασχολήθηκαν με τα πάντα εκτός από αυτά τα οποία αυτοί σε κάποια φάση είχαν προτείνει. Το πρόβλημα αυτό μέχρι τώρα δεν είχε ξεκαθαριστεί από πλευρά του Συμβουλίου. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει, θέλουμε να υπάρξει μια συζήτηση με το Συμβούλιο, να μας πει το Συμβούλιο τι αλλαγές προτείνει, να εκφραστεί πάνω στις αλλαγές αυτές το Κοινοβούλιο, να καταλήξουμε σε μία συνένεση, αλλά αυτή η σιωπή εδώ και δύο χρόνια του Συμβουλίου είναι μία ένοχη σιωπή και δημιουργεί προβλήματα στους Ευρωπαίους καταναλωτές και στις ευρωπαϊκές βιοτεχνίες. Λοιπόν, η Κυπριακή Προεδρία είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να το αγνοήσει και να πιέσει έτσι ώστε οι μεγάλες χώρες ε, αυτό που δεν έκαναν να το κάνει αυτή λόγω της αδιαφορίας για να μην πω ανικανότητας ορισμένων. Δεύτερο θέμα το θέμα του ΠΟΕ, των σχέσεών μας με τον ΠΟΕ. Γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχουν σημαντικές χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία που έχουν δώσει όπλα στη Συρία. Γιατί η Ρωσία, εδώ απ' έξω γίνεται και μια διαμαρτυρία, μια διαδήλωση, Η Ρωσία επίσης, η Κίνα μάλλον έχει καταπιέσει και καταστήλει με δύο τρόπο ε, τα Falun Dong ε, και γενικά παρόλα αυτά εξάγει στην Ευρώπη προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται από κρατουμένους οι οποίοι δεν έχουν δικαστεί ποτέ και δεν είναι προφανώς ένοχοι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν στην προσοχή του ΠΟΕ γιατί έτσι όπως είναι ο ΠΟΕ στη σημερινή φάση και έτσι όπως εργάζεται στην παρούσα φάση ο ΠΟΕ δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Η Αμερική σιωπά για δικούς της λόγους. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπως και η δική μου έχουν, που έχουν άμεσα συμφέροντα για εμπορικέ συμφωνίες με ορισμένες χώρες ή με ομάδες χωρών στον κόσμο με τον τρόπο αυτό δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες οι οποίες να μην παρέχουν ασφάλεια στις αγορές. Τέλος, μια δόση ελπίδας. Γνωρίζουμε ότι από το μήνα Αύγουστο επιτέλους στη Σομαλία θα υπάρχει ένας εκλεγμένος πρόεδρος. Μάλλον ο σημερινός πρωθυπουργός της Σομαλίας, ένας άνθρωπος ο οποίος την χάνει γενικής αναγνώρισης. Παρά τα άσχημα γεγονότα στην Κένια πρόσφατα, φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση επανελέγχου των τρομοκρατικών οργανώσεων στην Σομαλία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αρχή της διαδικασίας πολιτικής εξομάλυνσης στη χώρα αυτή. Έθεσα το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέτω και στο Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την δυνατότητα βοήθειας προς τη Σομαλία έτσι ώστε σε ορισμένα προϊόντα της να υπάρξουν διευκολύνσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την κατάσταση των πολιτών της χώρας αυτής, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχει μικρή φτώχεια υπάρχει και μικρή τρομοκρατία. Τελευταίοι ομιλητές και κλείνει ο κατάλογος. David Martin από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις ε, θέματα που έχουν ήδη αναφερθεί. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κέλλερ έθεσε το ζήτημα της άκτα και το τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε. Ε, μπορεί, αναρωτιέμαι αν το Συμβούλιο μπορεί να αντλήσει το δίδαγμα πως ε, η άκτα είναι νεκρή, την σκότωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Δεύτερον, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, συζητούσαμε τον κανονισμό πρόσβασης στην αγορά και ο μίλησε γενικά για τις συμφωνίες αυτές αλλά δέχεστε πως η προθεσμία της ε, Κομισιόν ε, για την απόσταση προτιμήσεων από χώρε την 1η 1 η 2014 δεν είναι ρεαλιστική και αυτό το οποίο προτείνει η Επιτροπή μας, δηλαδή 1η 1η-1η 2016 είναι πιο ρεαλιστικό. Τρίτο μου ερώτημα αφορά ιδιαίτερα την Ιαπωνία. Θα περιμένετε μέχρι το Κοινοβούλιο μας να συζητήσει τη διαπραγματευτική εντολή της ε, Ιαπωνίας πριν δώσει τη διαπραγματευτική εντολή στην Κομισιόν το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, David. Σύντομος και ουσιαστικός, όπως πρέπει. Ε, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω τον κύριο Υπουργό. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Μια γενική ερώτηση, η οποία είναι προφανώς, αναλαμβάνεται την ε, Προεδρία στο πέμπτο έτος της οικονομικής κρίσης και το εμπόριο έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει στο να βγούμε από την κρίση, αλλά εάν είναι εμπόριο που γίνεται ε, με την ίδια νεοφιλελεύθερη λογική που μας έφερε σε αυτό το χάλι δεν θα βοηθήσει τον κόσμο στην Ευρώπη ούτε αλλού στον κόσμο. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα διαφορετικό όραμα εμπορίου με βάση την αλληλεγγύη, αηφορία κτλ. Και δεύτερον συγκεκριμένα για την νότια γειτονία. Οπωσδήποτε η οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Παλαιτών έπαιξαν έναν έσχορο ρόλο στηρίζοντας ε, δικτάτορες στην περιοχή. Τώρα αυτοί που έκαναν τις επαναστάσεις στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, δικαίως είναι επιφυλακτικοί για τις προθέσεις της Ένωσης όταν ε, μιλάμε για διαπραγματεύσεις για το εμπόριο κτλ. Πώς θα καθησυχάσετε αυτούς τους ανθρώπους και θα οικοδομήσετε εμπορικές σχέσεις σε τελείως διαφορετική βάση, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, η περιφερειακή ολοκλήρωση κτλ. Και τελευταίο ερώτημα για την άκτα πάλι, η απάντησή σας, δηλαδή η προσέγγιση της Κομισιόν είναι σαφής, όπως λέει ο Ντέιβιντ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ξαναφέρει την άκτα, να συνεχιστεί η υπόθεση στο ΔΕΚ, και να επανέρχεται συνεχώς. Ε, θεωρούμε πως ε, εάν επανέλθει η Κομισιόν το Συμβούλιο πρέπει να αντιδράσει. Και τέλος κύριε Παδοπούλου, Σοσιαλδημοκράτη. Ε, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες δύο μέρες παρακολουθώ τους Κύπριους υπουργού να παρουσιάζουν τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές και περιορίζονται ακριβώ αυστηρά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και λένε ακριβώ τι προτεραιότητε που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Πριν από λίγο άκουσα μια ερώτηση και θέλω να διευκρινίσει ο κύριο Υπουργό. Μίλησε η κυρία Κέλλερ, άκουα τη μετάφραση στα ελληνικά, μίλησε για βορρά και νότο στην Κύπρο, αν μεταφράστηκε σωστά, και για την άμεση ανάγκη έναρξη απευθεία εσωτερικού εμπορίου ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αν να πρόκειται για δύο ξεχωριστά κράτη. Θα ήθελα να σχολιάσετε αν στην Κύπρο υπάρχει Βορράς και Νότος, δύο ξεχωριστά κράτη, ή ε, και τι γίνεται όσον αφορά τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων πολιτών. Πόσο αντιμετωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία όσον αφορά και το θέμα του απευθείας εμπορίου. Thank you very much for the question. ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας, ε, δεν μπορώ να σας δώσω απεριόριστο χρόνο για να απαντήσετε, αλλά δεν έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρώτα πρώτα να, να ξεκινήσω ε, από τα καλά λόγια ε, που είπε ο προφέσορ Μορέιρα και να σας πω ότι αυτά που αναφέρθηκε για την αρχή της Προεδρίας μας, αυτό είναι και ένα δείγμα της ε, εξαιρετικής δουλειάς που μπορεί να γίνει μέσα από τη συνεργασία του Συμβουλίου μαζί με το Κοινοβούλιο. Ε, και θεωρώ είναι σε αυτόν τον δρόμο που πρέπει να προχωρήσουμε. Όπως επίσης να πω κύριε Μωρέρα ότι είμαστε λίγοι στην Κύπρο αλλά ε, πρέπει να πω ότι έχουμε ανθρώπους λειτουργούς που δουλεύουν πάρα πολύ καλά, Κάνουμε εξαιρετική δουλειά έστω και αν είναι λίγοι γι' να αποδείχθηκαν ήδη από τις πρώτες μέρες της Προεδρίας μας και είναι πάνω σε αυτούς που στηρίζουμε και εμείς τη δουλειά μας. Τώρα έχουμε στα ε, ερωτήματα. Ήθελα να ξεκινήσω από το ε, ερώτημα του κύριου Κασπάρη ε, σε ό,τι αφορά τις χώρες της ΑΚΕ. Πρέπει να πω ότι η, η, η, η προτινόμενη τροποίηση του κανονισμού πρόσβαση στην αγορά δεν προτίθεται να αναγκάσει τι χώρε του να υπογράψουν συμφωνίε. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί τι δεσμεύσει που έλαβε, ανέλαβε όταν ο κανονισμό αυτό ε, τέθηκε ε, σε ισχύ. Ε, και άρα ε, είναι σε αυτήν την κατεύθυνση που πρέπει να προχωρήσουμε τα πράγματα ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν αυτέ οι συμφωνίε. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για την σουρ, ε, που έγινε και ερώτηματα και αν δεν κάνω λάθος από την κυρία Κέλλερ πρώτα πρώτα βεβαίω ε, ε, πέραν από τα προβλήματα που αναφέρθηκα και αφορά τη στάση της Αργεντινής βεβαίω υπάρχει θέμα μετά βεβαίω το ε, στην Παραγουάη για να μην αναφερθώ ότι υπάρχουν πάρα πολλέ άλλε δυσκολίε στο να προχωρήσουν αυτέ οι φωνίε δεν μπορεί, και αυτό είναι κανόνα, το είπα και στην εισαγωγή μου ε, παρέμβαση, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν απτύσσει εμπορικέ σχέσει δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι δημοκρατικέ ελευθερίε και πώ λειτουργούν σε κάθε ε, κράτο αυτό που θέλουμε να είναι εμπορικό μα εταίρο. Ε, νομίζω ότι ε, για τα θέματα της Ιαπωνίας και επειδή αυτό το ερώτημα μπήκε από μερικού ε, ευρωβουλευτέ ε, και από τον κύριο ε, Λάγκε και από τον κύριο Βιώσα, από τον κύριο Κασπάρη, να πω ότι το θέμα της η Ιαπωνία επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον και θέληση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και αποτελεί ένα θετικό παραγόντα. Και εμεί πρέπει βεβαίω και συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, ε, ε, τη θέση για το Κοινοβούλιο, θα πω μια γενικότερη θέση, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το ερώτημα, το, αυτό το θέμα το έθιξε και ο κύριος ε, Σούρτς. Ο κανονισμός είναι ότι ανατίθεται μια εντολή και όταν ολοκληρωθεί μια συμφωνία ερχόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Θεωρώ ότι υπάρχουν ε, αρκετοί τρόποι για να υπάρχει μια επαφή άτυπη, να μπορεί το Συμβούλιο και η Επιτροπή να ακούνε τι απόψει του Κοινοβουλίου πριν να καταλήξουν σε κάποιε συμφωνίε. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η αρχή μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι κάτι που το συζητήσαμε και με την αντιπροσωπεία τη ΙΤΑ όταν επισκέφθηκε την Κύπρο και τον κύριο, ε, τον κύριο Μορέιρα. Και νομίζω ότι αυτό Μπορεί να βρούμε τρόπου. Φτάνει να υπάρχει πολιτική βούληση ότι ω νομοθέτες πρέπει να βρίσκουμε του τρόπου για να εκφράζονται και να έχει υπόψη του το Συμβούλιο και η Επιτροπή τη του Κοινοβουλίου. Στην ε, ερώτημα του κύριου α, ε, Κασπάρη για τη ΣΥΠΑ, ε, συμφωνούμε πρώτα-πρώτα να πούμε ότι είναι γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η ΣΥΠΑ... Ε, έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο εμπορικό συναλλαγό στον κόσμο. Είναι δύο βασικοί εταίροι, είναι μια βασική μας ε, προτεραιότητα και ε, ε, με βάση την ενδιάμεση έκθεση που κυκλοφόρησε τη ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου για την απασχόληση και την ανάπτυξη στι 20 Ιουνίου, οι δύο πλευρέ είναι πρόθυμε να συνεργαστούν για ολοκλήρωση μια περιεκτική συμφωνία που να περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια της συμφωνία Ελευθέρων πορείων. Άρα είναι ένα θέμα που είναι στις προτεραιότητες μας. Ε, στα ερωτήματα του κυρίου α, Λάγκε, Yes, Διαδικαστικό, ναι κύριε Κασουλίδη, έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Κασουλίδη. Μικρόφωνο παρακαλούμε. να υπάρχει και μια αίτηση να μειώσετε την ταχύτητά σας γιατί η μετάφραση δεν απεικονίζει πλήρως αυτά τα οποία λέει ο κύριος Υπουργός ακόμα και στα ελληνικά και στα αγγλικά και μήπως θα μπορούσα να ζητήσω λέει ο πρόεδρος τον κύριο Σιλικιώτη να μειώσει την ταχύτητά του. Ε, στα ερωτήματα που ε, έθεσε ο κύριος Λάγκη Νομίζω ότι ε, ε, ε, για, την Ιαπωνία απάντησα. Τώρα για τι τις στρατηγικές κατευθύνσεις. να πω κύριε Λάγκη έχετε δίκιο. Στο σημερινό κόσμο με τα προβλήματα, τη μεγάλη κρίση που υπάρχει, τον μεγάλο ανταγωνισμό, η κρίση δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε μια περιοχή του είναι ένα θέμα που όλε οι πολιτικέ που στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλουμε πραγματικά να βγούμε από την ύφεση και να οδηγούμε στην ανάπτυξη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και το μοχλό του Διεθνού εμπορίου μαζί με όλα τα άλλα εργαλεία. Ε, Στι προηγούμενε μέρε στι επιτροπέ του Ευρωκοινοβουλίου συζητούσαμε για τα θέματα τη διεύρυνση τη αγορά, για τα θέματα τη βιομηχανία, για τα θέματα τη επιχειρηματικότητα. Δεν μπορούμε όλα αυτά να τα βλέπουμε ξεχωριστά ε, και να βλέπουμε πραγματικά ότι η εμπορική πολιτική είναι κάτι το αυτόνομο η εμπορική πολιτική είναι μέρος της πολιτικής για την ανάπτυξη που πρέπει ε, να ακολουθήσουμε και είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να αφήσουμε αυτή την ανάπτυξη. Ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που ε, θέσετε κύριε Λάγκε ε, σε σχέση με την Κίνα, ε, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν προβλήματα, όμως δεν μπορούμε να παραβλέπουμε το γεγονός ότι με την Κίνα μπορούμε να αναπτύξουμε σημαντικές εμπορικές σχέσεις. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι ε, ε, η προσπάθεια μας πρώτα είναι να ε, έχουμε μια επενδυτική συμφωνία χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα γίνει η συμφωνία χωρίς κανόνες και μέτρα και αρχές πάνω στι οποίες πρέπει να στηρίζεται το διεθνές εμπόριο. Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα του ε, κύριο Στάρτη. Ε, για τις προτεραιότητες νομίζω ότι ε, έχω αναφερθεί σε συμφωνίες. Δηλαδή ο Καναδάς βεβαίως θα ολοκληρωθεί, η Σιγκαπούρη, είμαστε σε ένα διάλογο καλά προχωρημένο με την Μαλαισία και βεβαίως έχουμε πρόθεση αυτό που ανάφερα να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και ε, να ολοκληρωθούν βεβαίως και οι συμφωνίες με τις ε, χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης, τη Γεωργία, την Αρμενία. Για την αποτελεσματική πολιτική εμπορίου, σε ό,τι αφορά τον εξυγχρονισμό και τα αμυντικά εργαλεία που αναφέρθηκε, κύριε Στάρτη, βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίζουμε το διεθνέ εμπόριο και εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα-πρώτα με μια σκοπιά περισσότερη φιλεύθερη. Εμεί ε, πολλέ φορέ ε, ε, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε μέτρα προστατευτισμού που αναλαμβάνουν άλλε χώρε. Άρα, χωρί τούτο να παραβλέπει το ότι πρέπει να θέτουμε συγκεκριμένα ζητήματα, εν η στόχη μας πρέπει να είναι να ενισχυθεί και το πολυμερές και το ε, διμερές εμπόριο. Ε, στα ερωτήματα που έθεσε η κυρία ε, Κέλλερ, ε, πρώτα πρώτα να πω, να ξεκινήσω από το θέμα της άκτα επειδή το θέσαν και άλλοι. Η Επιτροπή έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αναμένουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μετά όμως την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή η απόφαση το Συμβούλιο και η Επιτροπή να μην τη λάβουν υπόψη. Άρα ε, θεωρώ ότι έχουμε σήμερα νέο δεδομένο και στη βάση αυτού του δεδομένου πρέπει να λειτουργήσουμε σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα αυτά. Ε, για το θέμα της του απάντησα. Τώρα για την Κύπρο πρώτα πρώτα να πω ότι ε, Υπάρχει ένα ε, κυρία Κέλλη, ένας ε, κανονισμός εμπερού για την πράσινη γραμμή. Δεν είναι εμπόριο μεταξύ Κυπριακή Δημοκρατία και του Βορρά. Μέσα από αυτόν τον κανονισμό του εμπορίου διευκολύνονται οι τουρκοκύπροι πολίτε τη Κυπριακή Δημοκρατία ε, στο εμπόριο. Και είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Πέραν από αυτό το γεγονό, να πω ότι οι πολίτε τη Κυπριακή Δημοκρατία, και αναφέρομαι στου Τουρκοκύπριου, ανεξάρτητα διαμένουν στα κατεχόμενα, έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω ακόμα ότι ε, και στα νοσοκομεία έχουν πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαψη σε αντίθεση με τους ελληνοκύπριους που η πρόσβαση τους στα νοσοκομεία είναι στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων. Άρα θεωρώ ότι ε, αυτά όλα γίνονται ακριβώς γιατί λαμβάνουμε υπόψη ε, τα, και τα συμφέροντα των ίδιων ε, των Τουρκοκυπρίων. Όμως, στο ευρύτερο θέμα, και λυπούμε γιατί αναγκάζομαι ως Προεδρεύω του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλώ για την ε, πατρίδα μου, για την Κύπρο, όμως θα πω μια γενική αρχή που νομίζω όλοι πρέπει να έχουν υπόψη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην υλοποίηση, και έτσι είναι μέχρι σήμερα, στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και εμεί όλοι πρέπει να αποδούμε και το διεθνέ δικαίωμα να εφαρμόζεται, αλλά να εφαρμόζεται και το κοινοτικό κεκτημένο. Και είναι αυτό που είναι η απέτησή μα. Και εξάλλου νομίζω ότι ε, τα θέματα του ε, κανονισμού τα απευθεία ε, είναι ένα ζήτημα που πλέον υπάρχει μια ξεκάθαρη νομική βάση και νομίζω έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζω στη βάση αυτής της νομική βάσης, όπως επιτάσσει εξάλλου ε, τα ίδιες οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στα ερωτήματα του ε, κύριου Σούτς να πω ότι ε, του κύριου ε, εμείς πρώτα πρώτα να πούμε ότι στα θέματα του Τη κατάσταση που έχει να κάνει με τον γύρο τη Ντόχα. Ε, την ε, Επιτροπή. Είναι μια κατάσταση που ε, βρίσκεται σε τέρμα. αφού τα μέλη του ΠΟΕ δεν κατόρθωσαν μέχρι στιγμή να ολοκληρώσουν μεταξύ τους διαπραγματεύσεις. ωστόσο, η παρούσα φάση δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ω μια ενδιάμεση και μεταβατική αφού όλα τα μέλη του ΠΟΕ εξακολουθούν σε κάθε ευκαιρία να δηλώνουν την προσήλωσή του στην, σε μια θετική ε, κατάληξη. Στα θέματα του, του ΆΚΕ και του Συμβουλίου νομίζω ότι ε, εμείς ε, ε απάντησα προηγουμένως στα, σε αυτά τα ερωτήματα. Ε, στα ερωτήματα της κυρίας Μορκαντίνη να πω ότι η κυρία μοσκαρτινη ε, ε, πρώτα πρώτα ε, έθεσε κατά μου σωστά το θέμα σε σχέση με το εμπόριο που γίνεται. Είναι αυτό που απάντησα. για το γεγονός, για το φάκελο, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει από το Συμβούλιο να δημορφώσει τη θέση του προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Είναι γνωστό ότι όντω ότι υπάρχουν έντονε ανησυχίε σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών, οι οποίες πρέπει να γίνουν ε, σεβαστές. Παρά τις εντατικές προσπάθειες που έγιναν από προηγούμενες προεδρίες, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο υπέρ της πρότασης. Ε, η ιδέα της ε, εφαρμογής της, της ενός συστήματος σε εθελοντική βασή διερευνάται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτά όλα νομίζω θα βοηθήσουν ώστε ο κανονισμός προέλευσης των προϊόντων ε, να ε, προχωρήσει. Ε, ο κύριος Μάρτιν ε, Νομίζω για τα θέματα της τα απαντήσαμε, για τις, ε, ε για ε, εταιρικές ε, σχέσεις. νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να βρούμε, κύριε Μάρτη, μια συμβαστική λύση. Καταλαβαίνω αυτό που εννοείται, ότι αν είναι πιο ρεαλιστικό, όμως θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε μια συμβαστική λύση με το Ευρωκοινοβούλιο. Για την Ιαπωνία, ε, το Συμβούλιο ε, κανονικά πρέπει να περιμένει την άποψη του ε, Ευρωκοινοβουλίου. Ε, στα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Μάρφιν, ε, ε, πρώτα πρώτα να πω ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε τις σχέσεις με τις χώρες της περιοχής. Λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε τα ζητήματα ε, των ε, ε, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες. Πρέπει να βοηθήσουμε τη δημοκρατική διαδικασία που ξεκίνησε στις γειτονικέ μας χώρες. αντιλαμβάνουμε ότι μπορεί να υπάρχει το οποιοδήποτε θέμα από το παρελθόν. Βεβαίω να πω ότι ε, το θέτουμε και ως προτεραιότητα γιατί πέραν από ότι Κύπρος είναι μια μεσογειακή χώρα έχει άριστες σχέσεις ε, με τους ε, Άραβες γείτονές μας και θεωρώ ότι θα μπορούμε να συμβάλλουμε να ξεκινήσουν οι, οι διαπραγματεύσεις για αυτές τις, με αυτές τις χώρες που θεωρώ ότι είναι και σημαντικό και για τις ίδιες τις χώρες αυτές αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω αγαπητέ Πρόεδρε προσπάθησα ε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα μέσα στον χρόνο που μου δώσετε να απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσαν οι, οι κύριοι Ευρωβουλευτές. Uh, Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Οπωσδήποτε δεν θα είναι τελευταία φορά που θα έρθετε. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες ε, για να ανταλλάξουμε υπόψεις για τη Βόρεια Κύπρο. Να σας υπενθυμίσω πως θα παραπέμψουμε τον κανονισμό εμπορίου με την ε, Βόρεια Κύπρο. Και τέθη το ζήτημα του εάν είναι θέμα διεθνούς εμπορίου και ζητήσαμε οδηγίες από την διάσκεψη των Προέδρων και δεν έχουμε λάβει απάντηση ακόμα. Οπότε το ζήτημα έχει παγώσει εκεί. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή επιτυχία για την Προεδρία σας και συγχαρητήρια και πάλι και στον ε, εκπρόσωπό σας στην ε, Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, τον ε, κύριο Ρούσο. Ευχαριστώ πολύ. let's move to the next item. Πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι το σημείο 14. Παρακαλώ καθίστε στις θέσεις σας ή αποχωρήστε. time Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάω σοβαρά. Το επόμενο θέμα είναι η παρουσίαση μιας μελέτης για την οικονομική σημασία της προσχώρησης της ε, Ρωσίας στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ο Δ. Ρίτσαρτ Κόνολι θα παρουσιάσει αυτή τη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του, Κέντρου του Μπέρμιχαμ, το Κέντρο για Ρωσικές και Ανατολικοευρωπαϊκές Μελέτες. Αυτή η μελέτη είναι ήδη έντυπη, έχω ένα αντίτυπο εδώ μπροστά μου και νομίζω ότι έχει διανεμηθεί σε όλους σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν τον κύριο Κόνολη και έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την μελέτη σας. Είναι PowerPoint η παρουσίασή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, είμαι συνηθισμένος να έχω στις παρουσιάσεις μου ένα ακροατήριο 10 ατόμων από τους οποίους ορισμένοι κοιμούνται και έχω ένα σήμερα πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο. Θα προσπαθήσω όμως να παραμείνω σε επίπεδο απλό. Θα χρησιμοποιήσω τα εργαλεία του Economist ορισμένα τυποποιημένα στοιχεία τα οποία ίσως είναι η υπεραπλοποίηση της πραγματικότητας. Εάν έχετε όμως στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα μπορούμε να επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Τρία σημεία. Καταρχήν, ποιε είναι οι κύριες δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί από την ε, Ρωσία για την προσχώρηση στον ΠΟΕ και χθε, όπως ξέρετε η Δούμα της Ρωσίας κύρωσε την απόφαση προσχώρησης στον ΠΟΕ. Μέσα σε 30 μέρες λοιπόν υποχρεώνει τη Ρωσία να προσχωρήσει και επισήμως. Δεύτερον, θέλω να δω μερικά από τα κύρια οικονομικά, τα πιθανά και οικονομικά αποτελέσματα αυτής της προσχώρησης. Και τρίτον, θέλω να δω ποιε θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειε για την οικονομική μεταρρύθμιση στη Ρωσία στο μέλλον. <clears throat> Πρώτα απ' όλα, η Ρωσία, όπως συνήθως κάνουν οι χώρες όπως παίρνουν στον ΠΟΕ, έχει δεχτεί να μειώσει τους δασμούς σε βιομηχανικά και άλλα αγαθά. Δεν είναι μεγάλη αυτή η μείωση των δασμών, γιατί η Ρωσία έχει προχωρήσει αρκετά σε φιλελευθερωποίηση σε τελωνιακό επίπεδο τα τελευταία 10 και 15 χρόνια. Ίσως το πιο σημαντικό τμήμα των δεσμεύσεων ήταν η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών. Και αυτό θέλω να τονίσω ότι είναι ένα σημαντικό τομέα ενδιαφέροντο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλε χώρε οι οποίε μπορεί να ενδιαφερθούν να επενδύσουν ιδιαίτερα στη Ρωσία. Αυτέ λοιπόν είναι οι κύριε δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ρωσία. Ποια είναι τα πιθανά οικονομικά αποτελέσματα. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα είναι σχεδόν περιορισμένο ο αντίκτυπο βάσει ορισμένων οικονομικών μελετών που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε ένα οριζόντα 5 με 7 ετών, αν όλα πάνε καλά, θα προσθεθεί το 3,5% του ΑΕΠ στην οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας σε αυτό το χρονικό ε, διάστημα. Δεν είναι σε αιτήσιο επίπεδο, είναι 3,5% πάνω σε ένα χρονικό οριζόντα 5 με 7 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα είναι δραματικό αποτέλεσμα θα κάνει τη Ρωσία μια από τι πιο πλούσιε οικονομίε σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι περιορισμένε λοιπόν, περιορισμένα τα ωφέλη. Άμα δούμε από πού προέρχονται αυτά, 72% ε, αφορούν την άρση των εμπορίων στι ξένε άμεσε επενδύσει, τηλεπικοινωνίε, ε, τραπεζικό τομέα, ε, ασφάλειες και άλλε υπηρεσίε. Αυτό είναι το κύριο κομμάτι λοιπόν από όπου θα μπορούν να προέλθουν κέρδη για τη Ρωσία. Κάτι λιγότερο από 20%, 18% από χαμηλότερες τιμές και μεγαλύτερο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές. Και αυτά θα είναι κέρδη για τους Ρώσους καταναλωτές ουσιαστικά. <clears throat> και τέλος, μόνο 10% του κέρδους θα προέλθει από αυξανόμενη πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές για τους παραγωγούς της Ρωσίας. Με απλά λόγια δεν πρόκειται η Ρωσία να κατακλείσει τις ευρωπαϊκές αγορές με τα αγαθά, του, αγαθά της. Παράγει κυρίως η Ρωσία πρώτες ύλε, φυσικό αέριο και πετρέλαιο που ήδη εξάγεται ούτως ή άλλως. Και επομένως η αύξηση σε πρόσβαση της αγοράς δεν θα βελτιώσει ιδιαίτερα τα πράγματα για τη Ρωσία. Τώρα θα γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά. Είπαμε τα τρία τέταρτα σχεδόν του κέρδου θα είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση σε επενδύσει. Βλέπουμε όμω την σύγκριση τη Ρωσία με άλλε χώρε του ΩΣΑ και μη, του ΩΣΑ και δείχνουν τα φράγματα, τα εμπόδια στις άμεσες επενδύσεις. Είναι ακόμα πολύ σημαντικά τα εμπόδια για άμεσε ξένε επενδύσει στη Ρωσία. Επομένω, το αν η Ρωσία θα μπορέσει να πετύχει αυτό το κέρδο κατά 75% είναι αμφισβητήσιμο, όπω βλέπετε εδώ, η Ρωσία ίσως είναι η χειρότερη χώρα σε ό,τι αφορά τους φραγμούς για άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό. Επίσης η Ρωσία έχει, λάβει, έχει αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις, αλλά συγχρόνως είναι μια χώρα η οποία έχει μειωμένη διοικητική ικανότητα στο εσωτερικό της. Ακόμα λοιπόν και αν ο Βλαντίμιρ Πούτεν βγάζει ένα ουκάζε, μια, δηλαδή εντολή σε όλους να κάνουν κάτι, αυτά δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστούν από τη μια μέρα στην επόμενη. Ο χάρτης αυτός δείχνει την ε, πρόσβαση, μάλλον την διοικητική ικανότητα και βλέπουμε ότι η Ρωσία είναι από τις χαμηλότερες, από τις πιο αδύναμε χώρες σε ό,τι αφορά τη διοικητική ικανότητα, δηλαδή τη δυνατότητα να εφαρμοστούν οι κεντρικέ αποφάσει. Επομένω, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ρωσία ε, προ τον ΠΟΕ, θα είναι αρκετά δύσκολα για τη ρωσική κυβέρνηση να εφαρμόσει όλες αυτές τις ε, δεσμεύσεις. Για να συνοψίσω λοιπόν τον οικονομικό αντίκτυπο, αν σκεφτούμε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των δεσμεύσεων της Ρωσίας είναι αυτό που αφορά τις ξένες επενδύσεις. Για να το επιτύχει αυτό η Ρωσία πρέπει να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και την ικανότητα της κυβερνητικής μηχανής να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις. Για να γίνει κάτι τέτοιο όμως θα χρειαστεί να υπάρξει μια σημαντική προσπάθεια οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Από πού θα προέλθει λοιπόν αυτό. Η όθηση για μεταρρύθμιση έρχεται είτε από έξω και το είδαμε αυτό να μπορεί δυνητικά να προέλθει από την προσχώρηση στον ΠΟΕ, μπορεί να έρθει και από το εσωτερικό μια χώρα. Μια εσωτερική ελίτ, η ελίτ γύρω από τον Προύτιν και άλλου μπορούν να αποφασίσουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Μια αυξημένη οικονομική μεταρρύθμιση. Μπορεί να έρθει και εκ των κάτω, δηλαδή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από την κοινωνία των πολιτών κτλ. Και ας δούμε τώρα ποιες είναι οι προοπτικές για όλα αυτά αν θα έρθει από έξω η όθηση για τη μεταρρύθμιση. Ο χάρτης αυτής που είναι κάπως μπερδεμένο δείχνει τις βελτιώσεις στην οικονομική απόδοση των χωρών που έγιναν μέλη του ΠΟΕ τα τελευταία 20 χρόνια. Αν βλέπετε κάτι, βλέπετε ότι είναι περίπου τυχαίο το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που προέρχεται από την προσχώρηση στον ΠΟΕ. Για κάποιες χώρες βελτιώνεται η κατάσταση, για άλλες γίνεται χειρότερη. Επομένω, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι από μόνο, από μόνο της προσχώρησης στον ΠΟΕ θα αυξήσει τις προοπτικές για οικονομική μεταρρύθμιση στη Ρωσία. Δεύτερον, θα έρθει εκ των άνω. Μπορεί να έρθει από τη ρωσική ελίτ. Μέχρι στιγμής Υπήρξαν κάποιες ε, θετικές δηλώσεις της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια, αλλά βλέπουμε να υπάρχει τέτοια εκ των άνω όθηση όταν υπάρχει αυξημένο ανταγωνισμό. Αλλά στη Ρωσία μειώνεται ο ανταγωνισμό. Έχει αυξηθεί η υπερσυγκέντρωση στι ρωσικέ επιχειρήσει, στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχει αυξηθεί η ισχύ των κρατικών φορέων και το ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και άλλες άλλους νευραντικούς τομείς. Αν δούμε λοιπόν τη γενική εικόνα φαίνεται ότι οι ελίτ αντί να προωθούν περισσότερο ανταγωνισμό και περισσότερη αποκέντρωση υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συγκέντρωση. Υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση λοιπόν τη οικονομική εξουσία τα τελευταία χρόνια. Επομένω, οι προοπτικέ για να προέλθει κάποια τέτοια όθηση εκ των άνω είναι, είναι κάπως όχρη, δεν είναι ιδιαίτερα προφανής. Τέλος, θα έρθει μια τέτοια όθηση εκ των κάτω. Αν δείτε αυτό το γράφημα εδώ, μετράει στον άξονα τον κάθετο το εισόδημα κατά κεφαλή των χωρών, ενώ κάτω μετράται η ποιότητα της κοινωνικής τάξης σε μια χώρα, δηλαδή η καταπολέμηση της διαφθοράς, λογοδοξία, κράτος δικαίου κτλ. Και αυτό που βλέπετε είναι ότι για μια χώρα του εισοδήματος της Ρωσίας σε ένα μεσαίο επίπεδο είναι πολύ χαμηλή η ποιότητα της θεσμικής της τάξης. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται πολλές φορές για τη Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφθορά, δεν υπάρχει ένδειξη ότι είναι οικουμενικό το κράτος δικαίου. Το τονίζω αυτό <clears throat> γιατί λόγω του επίπεδου εισοδήματος της Ρωσίας θα περιμέναμε τη Ρωσία να αναπτυχθεί με γρήγορα βήματα σε ό,τι αφορά μια ποιοτική θεσμική μηχανή. Αλλά αυτό που είδαμε τα τελευταίου, τους τελευταίους μήνες μετά και τις θεματηρίες που έγιναν μετά την χρονιά στη Ρωσία και πριν από την χρονιά, και που κάποιες από τις οποίες διαματήριες συνεχίζονται ακόμα βλέπουμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη αίτηση για καλύτερη διακυβέρνηση από την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία και αυτά είναι τα πρώτα δείγματα μια στάση η οποία μπορεί να αναπτυχθεί εν καιρό και να υπάρξει μια αίτηση από τον κάτω να λειτουργήσει καλύτερα η ρωσική κυβέρνηση. Αυτό έχει συμβεί και σε άλλε χώρε οι οποίε στη συνέχεια έγιναν πιο πλούσιε. Αλλά αυτό χρειάζεται τυπικά ένα χρονικό διάστημα δεκαετιών. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε προ καλύτερη ποιότητα των θεσμών στα επόμενα 10 με 15 χρόνια, αλλά αυτό είναι ένα θέμα μέσω πρόθεσμο με μακροπρόθεσμο. Εν κατακλείδη, η προσχώρηση στον ΠΟΕ θα έχει μονάχα περιορισμένη οικονομική σημασία για τη Ρωσία και για την οικονομική ανάπτυξη και για να τονώσει τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Είναι κάτι το θετικό η προσχώρηση, δεν έχει πιστεύω αρνητικές πτυχές, αλλά δεν είναι ένας καταλήτης που θα αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ρωσία. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Όπως είπα, οποιαδήποτε πρόοδο, οποιοδήποτε κέρδο που μπορεί να επιτευχθεί, εξαρτάται από μια βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα και μια βελτίωση στη διοικητική ικανότητα του ρωσικού κράτου. Ουσιαστικά θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι μπορεί οι εντολέ εκ των άλλων να εφαρμόζονται. Και όλα εξαρτώνται, πολλά εξαρτώνται από το αν οι ρωσικέ ελίτ θέλουν να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτή και να τονώσουν το επιχειρηματικό κλίμα και την ικανότητα της διοικητικής μηχανής. Και τέλος, το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ακόμα και αν υπάρξουν αυτές τις θετικές αλλαγές, και όλα αυτά είναι οικοτολογίες προς το παρόν, στα επόμενα χρόνια ε, θα χρειαστούν 10 ή 20 χρόνια για να αλλάξουν τα πράγματα και να φτάσει η Ρωσία σε επίπεδο ε, διοικητικής ικανότητας μιας χώρας του ΟΣΑ, αλλά θα μπορούσαμε Αντίθετα, να περιμένουμε τα επόμενα 10 με 20 χρόνια να φτάσει η Ρωσία στο επίπεδο της Βραζιλίας, του Μεξικού και της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ικανότητα αυτή. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε περιορισμένοι στις προσδοκίες μας για την Τουρκία, για, για την Ρωσία για τα επόμενα χρόνια και μια τελική παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι πολλά από τα πράγματα που θα γίνουν στη Ρωσία θα εξαρτώνται από το πετρέλαιο, το κύριο εξαγωγικό προϊόν της Ρωσίας, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο, η πιο σημαντική παράμετρος για το μέλλον της Ρωσίας. Αν οι τιμές παραμείνουν εκεί που είναι, το κίνητρο για να υπάρξει μεταρρύθμιση θα είναι περιορισμένο, είτε εκ των άνω είτε εκ των κάτω. Αν μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη πίεση και από την ελίτ και από την κοινωνία των πολιτών γενικά. Επομένω, η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου τα επόμενα 10 με 20 χρόνια πιστεύω ότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση τη Ρωσία σε σχέση με την οικονομική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόνολη. Υπάρχει η ομάδα παρακολούθησης των ρωσικών υποθέσεων. Υπεύθυνο είναι ο κύριος Στέρντι, του δίνω το λόγο. Ρόμπερτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε για την τελευταία σας διαφάνεια με τα συμπεράσματά σας. Είναι πολύ νωρίς βέβαια γιατί η Ρωσία ε, μόλις υπέγραψε την ένταξή της στον ΠΟΕ. Θα ήθελα να πω ότι ίσως σε ένα χρόνο ή και σε δύο χρόνια θα μπορέσουμε να πούμε κάτι. Οι εκτιμήσεις σας βασίζονται στις πληροφορίες τις οποίες έχετε πάρει από άλλες χώρες που έχουν ενταχθεί στον ΠΟΕ ή πιστεύετε ότι η Ρωσία πράγματι δεν πρόκειται να ωφεληθεί ιδιαίτερα. Εγώ δεν μπορώ να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα, τα υπέρ και τα κατά είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Πιστεύετε εσείς ότι δεν θα υπάρξει βούληση από πλευράς των Ρώσων να ανοίξουν τις αγορές τους και να δημιουργηθεί μια κάποια οικονομική πειθαρχία. Θα ακολουθήσει μια σειρά ερωτήσεων παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Κούτας και αυτός μέλος της ομάδας που παρακολουθεί τις ρωσικές υποθέσεις. Θα ήθελα να χαιρετήσω την επικύρωση από την Ρωσική Δούμα της συμφωνίας με τον ΠΟΕ. Πιστεύω και <clears throat> το πιστεύω βαθύτατα ότι η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα διευκολύνει το εμπόριο μαζί της. Και νομίζω ότι η ένταξη αυτή θα οδηγήσει στην σύναψη συμφωνιών κοινών κανόνων Ε, γεγονότα όπως η απαγόρευση εισαγωγής ζών των ζώων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να μην υπάρξουν ε, στο μέλλον ξανά. Πρέπει να είναι υψηλά τα επίπεδα των σχέσεών μας με τη Ρωσία. Πρέπει να κλείσουμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων το κεφάλαιο για την ενέργεια, το θέμα της αμοιβαιότητας, της έλλειψης διακρίσεων, είναι θέματα στα οποία θα πρέπει να καταλήξουμε. Αυτή θα πρέπει να είναι η στόχη μας. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά η αίσθηση την οποία έχω και η ελπίδα την οποία έχω είναι ότι η ένταξη της Ρωσίας στον ΠΟΕ θα είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό τουλάχιστον για μας. Ευχαριστώ Τζόρτζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η μελέτη δείχνει με εντυπωσιακό τρόπο τις πιθανές εξελίξεις στη Ρωσία, στη Ρωσική Ομοσπονδία μετά από την ένταξη στον ΠΟΕ. Θα μπορούσατε ίσως όμως να μας δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες ε, για το ανθρώπινο δυναμικό, το εργατικό δυναμικό στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία. Γιατί αν οι φόβοι που έγιναν στη συζήτηση στη Ρωσική Δούμα αντικατοπτρίζουν τους φόβους στη Ρωσική κοινωνία για τις πιθανές ε, επιπτώσεις της ένταξης της χώρας αυτής στον ΠΟΕ. Απαιτείται να υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια όθηση προς την ένταξη αυτή. Ε, αυτό θα εξαρτηθεί και από το τι θα συμβεί στο εργατικό δυναμικό. Θα αλλάξει η κατάστασή του Υπάρχουν ερωτήσεις από τα υπόλοιπα μέλη, λέει ο Πρόεδρος. So no more questions. Dr. Connolly, the floor is again to... Υπάρχουν λοιπόν άλλες ερωτήσεις. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές, κύριε Κόνολη. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω με τη σειρά που έγινε, λέει ο κύριος Κόνολη. Αν κατάλαβα καλά, με ρωτήσατε το εάν υπάρχει βούληση στη Ρωσία θετικό αυτό το οποίο είπατε, ότι σωστό αυτό το οποίο είπατε, πως πράγματι η ψηφοφορία στην ε, Δούμα ήταν, ε, κρίθηκε με λίγες ψήφους. Και αν δεν είχε τόσο πολλές έδρες η Ενωμένη Ρωσία, δεν ξέρουμε αν θα περνούσε από τη Δούμα κάτι τέτοιο, γιατί υπήρχε μεγάλη αντιπολίτευση βεβαίως τη δρασία από το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και από άλλα αριστερά κόμματα, ακόμα και από αυτά τα οποία συνήθως συμπλέουν με την κυβέρνηση στη Δούμα. Συνήθως, αν υποβάλει κάτι στη Δούμα η ρωσική κυβέρνηση, περνάει. Και το ότι τώρα πέρασε οριακά, μας δείχνει πως υπήρχε μια αντίσταση στην κοινωνία και από ό,τι φαίνεται μόνο ένα τρίτο του πληθυσμού, σύμφωνα με πολύ έγκυρη δημοσκόπηση, υποστηρίζει την ένταξη στον ΠΟΕ. Βεβαίως η κυβέρνηση είναι συγκεντρωτική και δεν είναι πάντα ευαίσθητη στη φωνή της ρωσικής κοινωνίας, η οποία δεν είναι πεπισμένη για το μακροπρόθεσμο όφελος. Και πράγματι είναι ακόμα νωρίς. Ρωτήσατε το, που είναι τα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα στην την εμπειρία οικονομικών μεταρρυθμίσεων με άλλες χώρες, οι οικονομετρικές μελέτες που εξετάζουν τη δομή της ρωσικής οικονομίας και του εργατικού δυναμικού και του πώς θα επηρεάζονταν. Με απλά λόγια, οι τομείς οι οποίοι δεν θα πάνε πάρα πολύ καλά είναι αυτοί οι οποίοι προστατεύονται από επίσημα και ανεπίσημα εμπόδια στο εμπόριο και τις υπηρεσίες ειδικά τα πιο τα λιγότερο εξελιγμένα κομμάτια της βιομηχανίας τα οποία έχουν μεγάλη ένταση εργασίας όπως και η γεωργία είναι οι κλάδοι που αντιστέκονται στην ένταξη των ΠΟΕ αλλά αυτό το οποίο θα έλεγα ε, είναι πως στις τελευταίες ημέρες διαβάζοντας τον ρωσικό τύπο βλέπουμε τμήματα της ρωσικής διοίκησης που λένε στο λαό πώς με διάφορους ε, τρόπους θα σας προστατεύσουμε από την ένταξη στον ΠΟΕ. Λένε δε πως αυτό θα γίνει εντός των κανόνων του ΠΟΕ και το ελπίζουμε, αλλά αυτό το οποίο είπα είναι πως ε, με βάση τη μειωμένη διοικητική ικανότητα του ρωσικού κράτους θα εγώ θεωρώ πως θα υπάρχουν κάποια εμπόδια στο εμπόριο. Κάτι άλλο ε, για το ότι λέτε πως θα είναι θετικό. Συμφωνώ Δεν λέω πως ε, θα υπάρξει κάτι το οποίο θα γίνει μεσοπρόθεσμα, θα είναι κάτι το οποίο θα γίνει σταδιακά. Ε, πράγματι η ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά το πρόβλημα με την ενέργεια είναι πως το κεφάλαιο αυτό είναι πως η Ρωσία εδώ πέρα έχει όλους τους άσους στο μανίκι. Έχει, είναι μια χώρα η οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένη, μεγάλο μέρος του πετρελαϊκού τομέα είναι στα χέρια ιδιωτών σε αντίθεση ξέρω με τη Βενεζουέλα ή τη Σαουδική Αραβία ε, είναι 50-50 στη Ρωσία ο τομέα στα χέρια του ιδιωτικού τομέα οπότε είναι ήδη αρκετά ε, ανοιχτό ο κλάδος αυτός και ε, βλέπουμε πως ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές απαιτήσει και αυτό ισχύει και για τα νέα πετρελαϊκά αποθέματα που θα εκμεταλλευτούν οπότε ούτω ή άλλω θα είναι εταιρείε υψηλή ε, τεχνολογίας. Τώρα, το αν θα υπάρξει κάποια ενεργειακή χάρτα για να γίνει αυτό επισήμω είναι άλλο θέμα, αλλά στο μικρό επίπεδο θα δείτε ε, πω οι εταιρείε θα πηγαίνουν στη Ρωσία γιατί ακριβώς ε, υπάρχουν και οι δυσκολίες για την εξερεύνηση στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Τέλος, αναφερθήκατε στο εργατικό δυναμικό βλέπουμε σε μια διαφάνεια εδώ πέρα στην ε, σειρά την ε, δεύτερη από κάτω βλέπουμε το τι προβλέπεται ως αποτέλεσμα της ένταξης των ΠΟΕ. Είναι μια πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας σε, σε ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργαζόμενους. Και αυτό το οποίο λένε είναι πως καθώς θα έρχονται ξένες εταιρείες, ε, τηλεπικοινωνιακές ε, και λοιπές. Ε, το ειδικευμένο προσωπικό θα έχει καλύτερους μισθούς και θα μπορέσει να αγοράσει καλύτερα προϊόντα, αλλά λένε πως το ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό δεν θα υποφεληθεί όσον αφορά π.χ. καλύτερους μισθούς, θα υποφεληθεί λίγο από τη μείωση των δασμών από πλευρά κατανάλωσης ε, και θα μπορέσουν να αγοράσουν αγαθά ψηλότερης ποιότητας, αλλά σε γενικέ γραμμέ λένε πω όταν ενταχθεί η ΠΟΕ θα χάσουν οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρεσία. Αν δούμε γενικώ το παγκόσμιο εμπόριο, τι εξελίξει τι τελευταίε δεκαετίε, αυτό γίνεται στι ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, τι χώρε του ΟΣΑ, εποφελείται το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι χάνουν καθώς ε, η παραγωγή πηγαίνει σε χώρες χαμηλότερου κόστος. Αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μου στην ερώτηση. Δηλαδή τώρα η Ρωσία που εντάσσεται περισσότερο στη διεθνή κοινότητα θα ζήσει τα ίδια προβλήματα που ζούμε εμείς, πως δηλαδή η ανειδίκευτη εργασία δεν επωφελείται τόσο πολύ από το αυξημένο εμπόριο. Ελπίζω, ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κόνολη, που ήρθατε να μας παρουσιάσετε τη μελέτη σας. Και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης. Ε, έχει έρθει ο κύριος ε, Επίτροπος. Σας καλωσορίζω και πάλι αυτή τη φορά θα μιλήσει για την ενδιάμεση έκθεση για την ομάδα υψηλού επίπεδου ΙΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δουλειές και την Ανάπτυξη, η οποία συνεστάθη στην τελευταία σύνοδο κορυφής με τις ΙΠΑ τον Νοέμβριο υπό την συμπροεδρία του κυρίου Ντεχούχτ και του Ρον Κέρκ εκπροσώπου για το εμπόριο των ΙΠΑ. Αυτή εξ αρχής είχαν πει πως θα υπάρξει μια έκθεση τον Ιούνιο, ε, η οποία παρουσιάστηκε, γι' αυτό είστε εδώ. Ας ακούσουμε λοιπόν την αξιολόγηση της Κομισιόν για την ενδιάμεση αυτή έκθεση, η οποία κάνει μια προσωρινή σύσταση πως ε, η συνολική διμερής συμφωνία επενδύσεων έχει τις περισσότερες θανότητες για δουλειές και ανάπτυξη. Κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Έχετε τον λόγο. Και το μικρόφωνο σας είναι αυτό εκεί. You can, you can keep it. Here, here microphones are on the left. Ε, εδώ είναι στα αριστερά τα μικρόφωνα. Κάτι, υπάρχει μονίμως κάτι στα αριστερά. Ξέρετε κύριε Πρόεδρε, στο δείπνο το ψωμί είναι πάντα στα αριστερά. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που μπορώ να σας ενημερώσω σήμερα για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα και ιδιαίτερα για την ενδιάμεση έκθεση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας ενημερώσω και για την πρωτοβουλία για τις υπηρεσίες στη Γενέβη και αυτό θα το κάνω στο τέλος της παρέμβασής μου. Όλοι γνωρίζετε τη σημασία των εμπορικών σχέσεων με τη ΣΥΠΑ. Άνω του 1,8 δις σε καθημερινή βάση ανταλλάσσονται μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά φτάνουμε σε 2-3 και στις δύο περιφέρειες. Ε, σχεδόν το 50% του ΑΕΠ και το 1 τρίτο και άνω του 1 τρίτου του εμπορίου ελέγχεται θα έλεγα από τις δύο πλευρές ε, του Ατλαντικού. Αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ δεν έχουν προηγούμενο. Πολλά μπορεί να γίνουν ακόμα. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2011 στη συνάντηση κορυφής δημιουργήσαμε μια υψηλωτά του επίπεδου ομάδα εργασία για τις θέσεις απασχόλησης έτσι ώστε μέσω επενδύσεων και αύξησης των επενδύσεων να βελτιώσουμε την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Προεδρεύουν τη συγκεκριμένη αυτής ομάδας εργασίας ο γερουσιαστής Κέρκ και εγώ ο ίδιος και εξετάζουμε τις επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Στι 19 Ιουνίου υιοθετήσαμε την ενδιάμεση έκθεση στα πλαίσια της οποίας καταλήξαμε στο προσωρινό συμπέρασμα ότι μια συνολική συμφωνία η οποία θα καλύπτει τα θέματα των επενδύσεων για τη δημιουργία της απασχόλησης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τις περισσότερες από τις προτάσεις οι οποίες έγιναν. Οι προτάσεις αυτές σε πολιτικό επίπεδο επιτρέπεται να παρουσιαστούν σαν ένα συνολικό πακέτο. Η διαδικασία λοιπόν που ξεκίνησε από τη συνάντηση κορυφής προχώρησε προς τη σωστή κατεύθυνση παρά κάποιους δισταγμούς. Οι Αμερικανοί προτείνουν μια συνολική αντιμετώπιση και όχι μια σειρά επιμέρους συμφωνιών. Αυτό είναι συμβατό με τα συμφέροντά μας γιατί θεωρούμε ότι μια συνολική συμφωνία θα μας επιτρέψει να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα στα πλαίσια της επιθετικής προστασίας των συμφερόντων μας όπως τα θέματα των υπηρεσιών, τα θέματα των προμηθειών κτλ. Μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει το σύνολο των FTAs και δασμολογικές ρυθμίσεις και υπηρεσίες και επενδύσεις, προμήθειες δημόσιες, ε, προστασία της ιδιοκτησίας, εμπορικοί κανόνες για τους δασμούς, για όλα τα αγαθά. Βασικό στόχος είναι να καταργηθούν όλες οι επιβαρύσεις. Βέβαια θα υπάρχουν κάποια γεωργικά προϊόντα, τα οποία λόγω της ευαισθησίας τους θα υφίστανται μια ειδική μεταχείριση και θα υπάρξει κατάργηση των επιβαρύνσεων μετά από μια μακρά, ε, ίσως οικονομική περίοδο. η συμβατή εσωτερική ή μάλλον η περαιτέρω σύμβαση των ρυθμίσεών μας και στις δύο περιοχές ε, είναι βασικός στόχος της συμφωνίας. Σεβόμαστε τις παραδόσεις της κάθε πλευράς, σεβόμαστε το δικαίωμα της κάθε πλευράς ε, να νομοθετεί ανάλογα με το επίπεδο προστασίας το οποίο θεωρεί κατάλληλο. Πολύ μεγάλη σημασία έχει η πρόσκληση προς εμπλεκομένους να κάνουν προτάσεις ε, έτσι ώστε στα πλαίσια των εμπορικών ρυθμίσεων να καταργηθούν οι διαφορές. Έτσι λιέντουμε το έδαφος για ένα φιλόδοξο επίπεδο συμφωνίας διατλαντικής, αν και, ε, και αρκετά ρεαλιστικό. Και εδώ θέλω και τη δική σας υποστήριξη. Κάποια επίπεδα, κάποιες ρυθμίσεις σε επίπεδο υπηρεσιών σαν παράδειγμα, θα καθοριστούν στα πιο φιλόδοξα επίπεδα των συμφωνιών που έχουν μέχρι τώρα υπάρξει. Θέλουμε να προχωρήσουμε και σε επίπεδο απελευθέρωσης και σε επίπεδο προστασίας των επενδυτών, λαμβάνοντας σαν σημείο αναφοράς τα υψηλότερα επίπεδα απελευθέρωσης και προστασίας τα οποία έχουμε καταλήξει στα πλαίσια των επιμέρους εμπορικών συμφωνιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προστατεύσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να βελτιώσουν την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και τα πλαίσια της εθνικής μεταχείρισης της εμπορικής δραστηριότητας. Και το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κάτι το οποίο ε, θα λύσουμε από κοινού και εκεί όπου υπάρχουν κάποιες διαφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες θα ανοιχνεύσουμε τρόπους περαιτέρω σύγκλησης και βελτίωσης της επικοινωνίας. Τέλος, και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουμε στη διατύπωση υπερσύγχρονων κανόνων εμπορικών, από κοινού επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο νομίζουμε ότι θα είναι παράδειγμα και για τις τρίτες χώρες. Διευκόλυνση ας πούμε του εμπορίου, κανόνες του ανταγωνισμού, πρόσβαση στις πρώτες ύλες, ενέργεια, οριζόντιες διευκολύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιβάλλον. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι τομεί στους οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε. Στις 19 Ιουνίου, στα πλαίσια της συνάντησης στο Λοσκάμπος, οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων μας ζήτησαν να ολοκληρώσουμε σαν ομάδα εργασίας το ταχύτερο δυνατόν και να παραδώσουμε τα συμπεράσματά μας μέχρι το τέλος του χρόνου έτσι ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Ανάμεσα λοιπόν στην στιγμή που ζούμε τώρα και στην τελική απόφαση θα υπάρξει ίσως και μία ενδιάμεση έκθεση. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους τομείς τους οποίους θα καλύψει η ενδιάμεση συμφωνία, προετοιμάζοντας έτσι καλύτερα τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει αρκετά καλά και στα πλαίσια των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων. Ελπίζουμε να ξεκινήσουν γρήγορα οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική συμφωνία και ταυτόχρονα έχει ζητηθεί να υπάρξει μια μελέτη επιπτώσεων. Εμείς λοιπόν ελπίζουμε να ξεκινήσουμε τις επίσημες διαπραγματεύσεις στις αρχές του 2013 και να κλείσουμε στις αρχές του 2014. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο θέμα της συζήτησης για τις υπηρεσίες στα πλαίσια του ΠΟΕ. Ήδη ο εισηγητής κ. Ντεμαρτή σας ενημέρωσε για το θέμα αυτό το μήνα Μάιο. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά στις διερευνητικές συζητήσεις σε σχέση με μια πολυμερή ε, διαπραγμάτευση τις ε, υπηρεσίες με μια ομάδα περίπου 20 κρατών στην Γενέβη στα πλαίσια του ΠΟΕ. Στις 5 Ιουλίου υπήρξε ένα κοινό έγγραφο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τον τομέα των υπηρεσιών. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για μια πολυμερή συμφωνία η οποία βασίζεται στη Γενική Συμφωνία του ΓΚΑΤ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες και επίσης να αναπτυχθεί περισσότερο σε σχέση με την πρόσβαση στις αγορές και τους σχετικούς κανόνες. Εμείς υποστηρίζουμε την συνέχιση και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής του ΓΚΑΤ. Θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Μπορούμε έτσι να ανοίξουμε και την πόρτα για να υπάρχουν και άλλες χώρες του ΠΟΕ οι οποίες θα συμμετάσχουν, κυρίως αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες διαδραματίζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών, αλλά μέχρι στιγμές στάθηκαν διστακτικές να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη φιλελευθερωποίηση για τις υπηρεσίες. Για την Κομισιόν αυτή η πρωτοβουλία είναι μια ευκαιρία να προωθήσουμε τους στόχους φιλελευθερωποίησης του εμπορίου σε ε, υπηρεσίες που εμείς προωθούμε στο DDA. Και η, η στάση μας περιλαμβάνεται μέσα στη γενική μας προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις του DDA. Εμείς λοιπόν θα σας καθίσουμε ενήμερους και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Μουρέιρα. Έχετε δύο θέματα λοιπόν τα οποία παρουσιάσετε, το ένα είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και το άλλο το θέμα των διαπραγματεύσεων για τα, τις υπηρεσίες ή διερευνητικές τουλάχιστον συζητήσεις για μια δυνητική μελλοντική συμφωνία πολυμερούς χαρακτήρα για τις υπηρεσίες. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο διαφορετικά θέματα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα μέλη της ομάδος παρακολούθησης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και τα πολιτικά κόμματα θα μπορούσαν να διαλέξουν να δώσουν αντί των συντονιστών τα δικά τους, στα δικά τους μέλη της Ομάδος παρακολούθησης για το, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Κάσπαρη. Επιτροπέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας και βεβαίω για την προσήλωση που έχετε δείξει στον τομέα των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων. Είδα πως ε, οι δύο προκάτοχοί σας ε, το θεωρούσαν, το είχαν αυτό το θέμα έτσι, από παιδί. Εσείς όμως ασχοληθήκατε πάρα πολύ σοβαρά με αυτό και γιατί ρωτάω, το 2006 πριν από 6 χρόνια ζητήσαμε με ευρία πλειοψηφία από την Κομισιόν να έχει μια ολοκληρωμένη διατλαντική αγορά και οι προσπάθειες δεν ήταν ε, ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Πέρσι ζητήσαμε την στρατηγική για τις δουλειέ και την ανάπτυξη και χαίρομαι που επιτέλους υπάρχει κάποια πρόοδος. Ενώ με την κατάσταση στον κόσμο έχουν μετακινηθεί πάρα πολλά πράγματα στον τομέα του παγκοσμίου εμπορίου, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ έχουν συνειδητοποιήσει πως το βάρος μας στο παγκόσμιο εμπόριο επιδεινώνεται, όχι δραματικά, και πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε τις προδιαγραφές μας δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τεχνικές προδιαγραφές της οικονομικής τάξης. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μια διατλαντική εταιρική σχέση. Και αν δούμε αυτά τα οποία μας είπατε και πως προφανώς και η αμερικανική πλευρά αναγνωρίζει πως υπάρχει εδώ πέρα κάτι το οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, τότε λέω ανοιχτά, θα χαιρόμουν εάν ε, και η γενική σας διεύθυνση και εσείς ε, δίνετε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το θέμα τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να απογειωθεί, νομίζω, αυτό το αεροπλάνο. Τώρα, αν δεν φτάσει στην στρατόσφαιρα, όπως σε ορισμένες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, καλό θα ήταν να προσγειωθεί τουλάχιστον κάποτε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, και εντός της δικής σας της θητείας το αργότερο το 2014. Αυτό είναι φιλόδοξο. Έχουμε εννέα μήνες για προετοιμασία και μπορώ να πω πως εμείς θα στηρίξουμε μια τέτοια συμφωνία γιατί είναι προς το κοινό μας συμφέρον και για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν ε, πέρα από το εμπόριο. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και λοιπές προδιαγραφές όπου χρειαζόμαστε τους Αμερικανούς και έχουμε μεγάλο συμφέρον να επιτύχουμε. Και πραγματικά σας παρακαλώ ε, να παρεμβείτε εδώ πέρα και εάν και ο πρόεδρος μας ακολουθήσει αυτή την πρόταση, δηλαδή εάν διαπραγματευτούμε μια τέτοια συμφωνία με τις ΕΠΑ. Δηλαδή, όταν λέμε πώς χρειαζόμαστε αμοιβαία αναγνώριση, ρυθμιστικές προδιαγραφές κτλ. Θα πρέπει και γρήγορα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσουμε τις προδιαγραφές εκείνες, ώστε να περνάνε τα πράγματα αυτά τα οποία απαιτούνται τώρα, στη φάση της προετοιμασίας έτσι ώστε στο τέλος να μην αποτύχει η εφαρμογή της συμφωνίας το ότι εμείς ασχολούμαστε με κανόνες οι οποίοι είτε είναι βλακώδεις είτε αφορούν μόνο την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν κύριε Πρόεδρε να φροντίσουμε η Επιτροπή μας μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, μεταφορών, ε, βιομηχανίας Γεωργίας, ναι, τουλάχιστον αυτές τις τέσσερις επιτροπές. να ε, τοποθετηθούμε θεσμικά και να βοηθήσουμε την Κομισιόν για τυχόν προβλήματα. Και για το δεύτερο θέμα των υπηρεσιών θα ήθελα να μας παρουσιάσετε κύριε Επίτροπε. Μιλήστε για 20 χώρες οι οποίες διαπραγματεύονται να μας εξηγήσετε γιατί το πώς δηλαδή θα υπάρξει η δυνατότητα μιας συμφωνίας ε, εντός του ΠΟΕ αλλά και εντός του πολυμερούς πλαισίου γιατί δυστυχώς δεν το κάνουμε αυτό αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, οπωσδήποτε. Νομίζω πως ε, εφόσον ένα σημαντικό κομμάτι αφορά τα ρυθμιστικά ζητήματα, σημαντικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να εμπλέξουμε και τις επιτροπές εκείνες οι οποίες είναι αρμόδιες για την εσωτερική αγορά, τις μεταφορές, ε, περιβάλλον κτλ. Επίσης να σας υπενθυμίσω γιατί το ξέχασα πώς αποφασίσαμε στην Επιτροπή μας να ξεκινήσουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τις ε, σχέσεις τις εμπορικές ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό επευκαιρία της έκδοσης της ενδιάμεσης ε, έκθεσης. Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο χρονοδιαγράμματος. 17-18 Σεπτεμβρίου θα δούμε το σχέδιο έκθεσης. Σεπτεμβρίου είναι οι προθεσμοί για τροπολογίες. Οκτώβριο σχέδιο έκθεσης, Ολομέλεια Οκτωβρίου, ψηφοφορία στην Ολομέλεια και σκοπεύουμε να έχουμε κάποιο λόγο στην ε, αρχική αυτή φάση και να εκφράσει από στο Κοινοβούλιο πριν ε, ε, συνέλθει η ομάδα εργασίας ΙΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, υποβάλει έκθεση στο τέλος του έτους. Εγώ θα είμαι ο είμαι και μόνο ο για την ομάδα παρακολούθησης. Σοσιαλδημοκράτης Μπεντ Λάγκε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σωστό είναι το ότι επιτέλους έχουμε μία προσέγγιση για μία συμφωνία τερικής σχέσης με τη ΣΥΠΑ. Βεβαίως ε, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Έχουμε πολλές εμπειρίες σε προσπάθειες που έχουμε κάνει για μια συμφωνία για μικρά και μεγάλα θέματα. Και πρέπει βεβαίως να δούμε πού θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Γιατί πέρα από το ζήτημα της ε, νομοθεσίας βεβαίως που πρέπει να δούμε, υπάρχει και το ζήτημα του χρονικού περιθωρίου. Έρατε πως μπορούμε οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις μετά τις προεδρικές εκλογές της ΕΠΑ και ένα εξάμεινο επίσης πριν από τις εκλογές του Κογκρέσου ξέρουμε πως δεν είναι δυνατή η διαπραγμάτευση οπότε έχουμε ένα παράθυρο 1,5 ε, έτους και πρέπει άρα να οριστούν κάποιες προτεραιότητες γιατί Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να ε, κάνουμε τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού θα δώσουμε βάρος. Στους δασμούς ε, υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ μικροί δασμοί. Υπάρχουν ε, τομείς όπου είναι πολύ ψηλοί δασμοί. Π.χ. στα φορτηγά. Πάνω από 20%. Οπότε και στους δασμούς να δούμε πού είναι τα στρατηγικά μας συμφέροντα. Και στα μη δασμολογικά ζητήματα. Παρακολούθησα τη διαπραγμάτευση για έναν κοινό κύκλο μέτρησης εκπομπών φορτηγών. Εδώ και δεκαετίες παρακολουθώ αυτή τη διαδικασία και βλέπω πως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί ξανά και ξανά υπάρχουν ζητήματα ανταγωνισμού. Οπότε σας παρακαλώ να δούμε και τα μη δασμολογικά ζητήματα έτσι ώστε το πακέτο αυτό να μην είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και να έχουμε και κάποιο ρεαλιστικό τέλος. Ε, Aldi Group. Η ομάδα των φιλελευθέρων. Ο Ρόμπερτ Στέρτη έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ, όπως είπε ο Ντάνιελ, εντυπωσιάστηκα θετικά από την προσέγγισή σας. Χωρίς μικρόφωνο παρέμβαση. Εγώ φταίω, εγώ φταίω. Η Μαρή και είναι παρούσα και είναι μέλος της ομάδας παρακολούθησης, οπότε θα πάρει αυτή η πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αν θα κάνετε πρώτα τους συντονιστές και μετά τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Είμαι μέλος και της αντιπροσωπείας με τις ΗΠΑ και ασχολούμαι με διάφορες ιδιότητες με τις διατλαντικές σχέσεις. Θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα, γιατί πολλά έχουν ήδη αναφερθεί στην ενδιάμεση έκθεση και με αυτά που είπαν οι άλλοι συνάδελφοι. Θέλω να σταθώ στις ευκαιρίες να υπάρξει προτυποποίηση για τις τεχνολογίες και αντιμετώπιση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το τομέα εμπορίου τι προοπτικές βλέπετε και κάπως γενικότερα ποιος περιμένει ότι θα μπορούσε να είναι ο αντίκτυπος των σχέσεων μεταξύ της ε, σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεών μας με τρίτες χώρες στρατηγικά σε ό,τι αφορά το εμπόριο, παραδείγματος χάρη με την Κίνα, με άλλες αναδυόμενες ε, οικονομίες, όταν βελτιωθεί η σχέση μας σε εμπορικό επίπεδο με την, ε, τις Πολιτείες. Ο συντονιστής λοιπόν και των Πρασίνων και μέλος της ομάδας παρακολούθησης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, είναι μεγάλη χαρά να σας βλέπουμε μεταξύ μας. Αναφερθήκατε σε ένα αεροπλάνο. Ο Ντάνιελ αναφέρθηκε σε ένα αεροπλάνο. Ένα τέτοιο αεροπλάνο που πάει πολύ γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε είναι το Concorde. Αλλά στην τελευταία του πτήση το Concorde έκανε το πολύ 25 χιλιόμετρα και μετά έπεσε. Επομένως ίσως δεν είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα η προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Εδώ θα ήθελα να καταλάβω το εξής. Πέραν των πολιτικών δηλώσεων και προθέσεων, ποια είναι η πραγματικότητα, πού βρισκόμαστε σε σχέση με την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών που θέλουν να έχουν μια ενιαία διαπραγμάτευση και των Αμερικανών που θέλουν κατατομής διαπραγματεύσεις. Έχουμε καταλήξει κάποια συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις και η συμφωνία, τη μορφή της συμφωνίας που επιζητούμε επίσης. <clears throat> Εφόσον μας ενδιαφέρουν κυρίως τα κανονιστικά θέματα, εγώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσέγγιση στα συστήματα πιστοποίησης. Αλλά υπάρχουν και θέματα που είναι επαχθή, δύσκολα, η γεωγραφική προέλευση, οι πολιτιστικές, ε, ιδίω οι, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη Γαλλία, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τα θέματα χρήση ορμονών ή όχι στο βόλιο κρέα, μπορεί κανεί να απαριθμίσει πάρα πολλά θέματα όπου θα δει τελικά ότι για αυτά τα θέματα κανονιστικά, τα θέματα ρυθμίσεων, δεν πρόκειται μονάχα μη δασμολογικά εμπόδια. Μπορεί να μιλήσουμε περισσότερο και καλύτερα για συλλογικές προτιμήσεις και είδα ποια είναι η στάση του ΕΛΚ για τα θέματα αυτά. Επειδή θα έχουμε πολλά προβλήματα σε κανονιστικό επίπεδο με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μειώσουμε δυνητικά τουλάχιστον το κανονιστικό μας πλαίσιο για να είναι πιο εύκολη η διαπραγματεύση. Αλλά αυτό δεν είναι η οδηγός γραμμή της Ευρώπης, γιατί όπως έλεγε ο Μπεντ Λάγκε για τα φορτηγά, για τα καμιόνια, έχουμε και άλλα διακυβευόμενα, παραδείγματος χάρη εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος τα αμερικάνικα καμιόνια αν έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αυτό δεν μπορεί να γίνει αμέσως. Έχουμε λοιπόν κοινωνικού χαρακτήρα θέματα για τα οποία έχουμε βαθιές διαφορές με την ε, Αμερική και αυτό ξεπερνάει απλώς τις ε, εμπορικές διαφορές ή διαφορές για τα θέματα γεωργίας. Χρειάζεται και πάλι να υπάρχει μια πολιτική θέληση και είναι θεμητό να επιζητούμε μεγαλύτερη συνεργασία με τις ΗΠΑ αλλά Πώς θα αντιμετωπίσετε εσείς όλα αυτά τα προβλήματα που ξεπερνούν το στενά εμπορικό τομέα και ποιες προοπτικές έχετε. Και ένα τελευταίο σημείο, επειδή μιλήσατε για τις διαπραγματεύσεις και τις υπηρεσίες των ΠΟΕ, το γεγονός ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται δυνητικά μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, τι σημαίνει αυτό για τις πολυμερείς προοπτικές. Όταν υπάρχει μια, μια διαπραγμάτευση με τον Καναδά ή την Ιαπωνία ή τις ΗΠΑ, το γεγονός ότι τα μεγάλα εμπορικά μπλοκ όταν θέλουν να έχουν διαπραγματεύσεις μέσα στον ΠΟΕ για να έχουν κανόνες, τι γίνεται αν τελικά γίνονται σε διμέρες επίπεδο όλες οι διαπραγματεύσεις. Ο Ρόμπερτ Στέρθι, ο οποίος είναι όχι μόνο συντονιστής των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, αλλά και μέλος της ομάδας παρακολούθησης της ΗΠΑ. Με με ευχαρίστησαν ιδιαίτερα αυτά τα οποία είπατε, εκτός από μία λέξη. Η λέξη αυτή είναι η λέξη που προκαλεί προβλήματα, γεωργία. Κάθε φορά που μιλάμε για γεωργία, ξαφνικά θα μιλήσω για εγκεφαλοπάθεια των βοηδών και για τις υπόλοιπες ασθένειες ε, των ζώων, <clears throat> τις ορμόνες κτλ. Όλα αυτά τα θέματα παρουσιάζονται και καταστρέφουν τις διαπραγματεύσεις. Λέω συστηματικά μπορούμε να περιθωριοποιήσουμε λίγο τη γεωργία. Ας τη βάλουμε λίγο στην άκρη. Είναι ξεχαριστό θέμα η γεωργία. Έχουμε πάρα πολλά να κερδίσουμε με μέσω μια συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ. Ας αγνοήσουμε λίγο τη γεωργία. Θα ήθελα την άποψή σας τώρα για τις εκλογές. πώς αυτές οι προεδρικές εκλογές θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις. Αναφερθήκατε επίσης στο χρονοδιάγραμμα των 18 ε, μηνών ουσιαστικά. Πάρα πολύ θετικό το βλέπω. Και τι γίνεται με την συμφωνία την εμπορική με τις χώρες του Ειρηνικού ωκεανού, στη λεκάνη του Ειρηνικού. Αυτό πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις μαζί μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε. Η έκθεση αναφέρεται σε ορισμένες πολλά υποσχόμενες ρυθμίσεις και πρότυπα. Δεν πρόκειται λοιπόν για, μόνο για αυτά. Ο στόχος είναι να έχουμε και μία συμφωνία ελευθερών εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ τίθεται και το θέμα πρώτων υλών. Στην Κοπεχάγη φάνηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να μπορέσουμε να φέρουμε τα θέματα αυτά διότι επέκυντο οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες του Κογκρέσου και οι βουλευτές φοβόντουσαν ότι αν τεθεί το θέμα αυτό των θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σωστά κάτω από τέτοιες συνθήκες. Πώς λοιπόν κατά την άποψή σα, αυτή η κοινή ομάδα εργασία θα πρέπει να λειτουργήσει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και να εξασφαλίσει ότι θα μπορέσει να γίνει με έναν τρόπο διάφανο αυτή η διαδικασία. Πώς θα πρέπει να συγκροτηθεί λοιπόν το θέμα αυτό των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων ε, οικονομικών εταίρων πώς θα εξασφαλίσει θέσεις εργασίας, οικολογική προοπτική, κοινωνική συμπερίληψη. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να τα επιτύχουμε όλα αυτά, ώστε να έχουν μια σχέση παραγωγική και καρποφόρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και όχι απλώς να επαναλθούμε μονάχα στη μεθοδολογία της ε, φιλελευθερωποίησης, η οποία οδηγεί σε απώλεια θέσεων απασχόλησης. Αν δούμε την πραγματικότητα την οικονομική και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα ήταν αποτυχημένες προσπάθειες. Η Κομισιόν επίσης το έργο της έχει ε, τονίσει βέβαια ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου σημαίνει έλλειψη ε, επικάλυψη σε οικονομικές ε, δραστηριότητες. Χάνονται βέβαια κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Αυτό Όμω δεν πρόκειται να αλλάξει σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Αν λοιπόν ε, δούμε το τωρινό χρονικό ορίζοντα και μίλησε ο κ. Κασπάρ για μια περαιτέρω επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών, δεν πρόκειται και παρόλα αυτά να προκύψει κάποιο αποτέλεσμα θετικό για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Και έρχομαι τώρα στα αγροτικά θέματα. Βέβαια είναι σημαντικό να ανοίξει η αγορά των ΗΠΑ για τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα αυτά. Είναι καυτά θέματα τα οποία πάρα πολλές φορές συζητούνται. Πιστεύω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα στις συζητήσεις αυτές και να προχωρήσουμε στο ταχύτερο δυνατό σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κατεύθυνση αυτή. Δεν αναφέρεται επίσης στην ενδιάμεση έκθεση καμία μνήμα για, την, ε, ε, κοινή, για, την, για ε, κοινές ερευνητικές προσπάθειες, για, την, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημόσιοι τομείς και στις, οι δημόσιες προμήθειες και στους δύο τομείς, στις δύο χώρες, συγγνώμη, χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην πολιτική μας, όπως τόνισε ο κύριος Κασπάρη, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λοιπόν, εμείς θα θέλαμε κάτι τέτοιο, μπορούμε να περιμένουμε ότι εσείς ως Επίτροπος και οι άλλοι Επίτροπε με τους οποίους θα πρέπει να συνεννοηθείτε, ότι μπορούμε να περιμένουμε ότι θα δώσετε μια μεγαλύτερη διαφάνεια στις προσπάθειές σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να έχει μια καλύτερη πληροφορία ώστε να μπορέσει να συμβάλλει κάπως πιο επικοδομητικά στα θέματα αυτά. Μετά από τη διάσκεψη κορυφής του Ιουλίου θα θέλαμε να ξέρουμε κατά πόσο το Συμβούλιο μπορεί να σκεφτεί λίγο περισσότερο και να προχωρήσει από την ενδιάμεση έκθεση σε μια τελική έκθεση. Now, other members of this... Λοιπόν, τώρα, τα μέλη της Επιτροπής μας, ε, Παύλο από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Δυστυχώς δεν μπόρεσα δεν θα μπορούσα, συγγνώμη, να ήμουν περισσότερο σύμφωνος μαζί σας σε σχέση με τη συμφωνία που επέχει το εμπόριο για τη δημιουργία πλούτου, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για τη δυνατότητα να βοηθήσει στην έξοδο από την κρίση που μαστίζει σήμερα την Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να επενέσουμε τις προσπάθειες που καταβάλει η Κομισιόν για να γίνει η διαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών ελευθέρου εμπορίου και συμφωνίες εταιρι... ε η συμφωνία με την Συνωμένες Πολιτείες και την Αμερικανική Ήπειρο, τα θέματα κοινών αξιών και κοινών στόχων. Εμείς συμμεριζόμαστε την ιδέα του να προωθήσουμε το ελεύθερο εμπόριο μέσα στις περιοχές μας, οι δύο αυτές ε, μεγάλες ενότητες, και αυτό όπως φάνηκε με την ναύτα, με την κάφτα και η θελάκ, η ενιαία αγορά της Λαρνικής Αμερικής, όπως φάνηκε και από τις διάφορες συμφωνίες που συνήψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Μεξικό, την ε, Χιλή και αυτές που επίκυνται με την Κολομβία, το Περού κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια φιλόδοξη αντιμετώπιση. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς βλέπει η Κομισιόν τη δυνατότητα σε ένα κοντινό μέλλον να υπάρχει μια ενσωματωμένη και ολοκληρωμένη ζώνη ελευθερών εμπορίου που να περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική. Από τους σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Ντεζίρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι αυτή η εικόνα ενός ολοκληρωμένου τρόπου λειτουργίας της διατλαντικής αγοράς, μιας μεγάλης ενοποιημένης αγοράς, είναι ένα όνειρο. Από την άλλη όμως αυτό άπτεται της αυτονομίας και των διακανονισμών, των διοικητικών, των περιβαλλοντικών, στον τομέα της υγιεινής, στον τομέα της γεωργίας. Υπάρχουν διαφορές και όταν βλέπουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα των φορτηγών που το έθεσε ο Λάγκε, όχι μόνο υπάρχουν διαφορές στον τομέα των εκπομπών, αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό κατά τομέα και κατά προϊόν, ποια είναι και τα οικονομικά αποτελέσματα γιατί πράγματι οι δασμοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί, οπότε το κόστος θα ήταν περιθωριακό σε επίπεδο εισόδων, γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάμε για τους πιο μεγάλους οικονομικούς εταίρους στον κόσμο. Δεν υπάρχουν λοιπόν εμπόδια ουσιαστικά, όμως στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια επιμέρους εμπόδια, αν τα καταργήσουμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι επιπτώσεις θα υπάρξουν στις βιομηχανίες, στην απασχόληση και στις δύο πλευρές. Θα ήθελα να μας πείτε επίσης ε, τι γίνεται και με την εμπορική συμφωνία την Αμερικανική, την Αλενά όπως λέγεται στα γαλλικά. Προφανώς ο Καναδάς είναι πολύ προχωρημένος και οι κανόνες που ισχύουν εκεί στο τομέα του περιβάλλοντος, ε, του εργατικού δυναμικού είναι συγκρίσιμοι, αλλά με το Μεξικό υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όταν τέθηκε σε λειτουργία η εμπορική συμφωνία Καναδά-Ευρωπαϊκής ε, <clears throat> συγγνώμη, Ηνωμένων Πολιτειών και Μεξικού δημιουργήθηκαν προβλήματα. προβλήματα. Και ε, τι θα γίνει με τα προϊόντα από το Μεξικό, σαν παράδειγμα, αν περνάνε από τις Ηνωμένε Πολιτείες θα μπαίνουν χωρίς δασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι θα πρέπει να μείνουμε σε κάποιους κανόνες οι οποίες είναι σε συγκεκριμένη φάση. Ε, αυτό είναι σαν στόχος. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα. Ε, κάνατε αναφορά στο γύρο της Ντόχας. Η βασική αρχή ήταν ότι δεν θα υπήρχε απόλυτη αμοιβαιότητα ανάμεσα στις ε, εκβιομηχανισμένες χώρες και στις υποανάπτυξη χώρες. Για τις υπηρεσίες ισχύει αυτό, γιατί εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Για τις δημόσιες προμήθειες, σαν παράδειγμα, η θέση σας είναι να απαιτήσετε την αμοιβαιότητα για να καλύψετε το θέμα των ε, δημοσίων προμηθειών στις αναδιόμενες χώρες. Και υπάρχει και ένας τομέας ε, για ειδικό. Μιλάμε για τις δημόσιες προμήθειες. Στη Γενική Συμφωνία υπάρχουν κάποιες ρήτρε οι οποίες ε, δεν μπορεί να λειτουργήσουν αναδρομικά για την προστασία των επενδυτών στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών κτλ. Υπάρχουν θέματα λοιπόν εδώ, θα πρέπει να δούμε πως ε, υπάρχει και χώρος εγγύησης για τις εθνικές πολιτικές. Γιατί αν έχουμε μία πολυμερή συμφωνία, της οποίας μία από τις συνέπειες είναι ότι οι τοπικές αρχές είναι απολύτως δεσμευμένες από εξ αρχής ανηλυμένες αποχρεώσεις απέναντι στις πολυεθνικές, τότε τα προβλήματα θα είναι πολιτικά και σοβαρά. Τώρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, είναι πολύ φιλόδοξη και σημαντική η υπόθεση αυτή και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν ανάπτυξη. Είναι όμως το θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους οι οποίοι υπογράμμισαν ότι ο γεωργικός τομέας και γενικότερα ο αγροτροφημικός τομέας θα έλεγα εγώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, ξεχωριστά. Πρόκειται για έναν τομέα στα πλαίσια των οποίων οι διαφορές μας και αναφέρομαι στις διαφορές ΙΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ μεγάλες. Γενετικά τροποποιημένα, ε, η ανατροφή των ε, γαλακτοφόρων ζώων, Έχουμε πάρα πολλές διαφορές, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε ότι έχουν απογορεύσει στις Ηνωμένε Πολιτείε, σαν παράδειγμα, την επεξεργασία και την κατανάλωση ε, κρέατος από άλογα. Ε, ε, στην Ευρώπη κάτι τέτοιο επιτρέπεται σε πολλές χώρες. Λοιπόν, έχουμε διαφορές, ιδιαίτερα σε μία φάση κατά την οποία εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τα προβλήματα που τίθενται και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι στην προσπάθεια αυτή. Εγώ σίγουρα θέλω ένα φιλόδοξο μεγάλο πρόγραμμα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά. Σαν παράδειγμα την λεγόμενη τριμερή εν πάση περιπτώσει προέλευση προϊόντων, δηλαδή προϊόντα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν συμφωνίες και που θα φτάνουν με μηδενικούς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται ένα θέμα εδώ λοιπόν. Τίθεται ένα θέμα με τη συμφωνία τη συγκεκριμένη οι νόμοι που υπάρχουν από πολύ παλιά στις Ηνωμένε Πολιτείες και επιβάλλουν την ονομασία προέλευση σαν παράδειγμα, στις Ηνωμένε Πολιτείες Για μας δεν ισχύουν. Ή σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά θα αντιμετωπιστούν με βάση την αρχή της αμοιβαιότητα, οπότε οι Ηνωμένε Πολιτείες μπορεί να μας αποστέλουν προϊόντα, αλλά θα πρέπει να βάζουν στο προϊόν αυτόν την ονομασία προέλευσης. Αυτά είναι επιμέρους θέματα λέγω, τα οποία όμως πρέπει καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Οι συνάδελφοι με πολύ συγκεκριμένο τρόπο νομίζω ότι μας μετέφεραν μία σειρά από παρατηρήσεων σημαντικών υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτού του προγράμματος. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να προχωρήσουμε σταδιακά, να εντοπίσουμε τους τομείς όπου πράγματι υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε άμεσα να αποφύγουμε να εμπλακούμε στα πλαίσια μιας κατάστασης που δεν θα προσφέρει εξόδους διαφυγής και να διευκρινίσουμε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα επιμέρους θέματα πριν προχωρήσουμε και στον τομέα της αμοιβαιότητας και στον, το, στο πιστοποιητικό προέλευσης και στο θέμα των προϊόντων που περνούν από τρίτες χώρες. Όλα αυτά είναι θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ. Δεν θα δεχτούμε άλλες ομιλητές. Η κυρία Άντρης από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που αυτή τη φορά μου επιτρέπετε να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Επίτροπο. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο από το 1989 η υπηρεσία του προσώπου για το εμπόριο των ΗΠΑ έχει λεγόμενη έκθεση 301 για το πλαίσιο πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων χωρών και μπορεί αυτές να υποστούν αντίπεινα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι να ικανοποιηθεί ο εκπρόσωπος πως υπάρχει επαρκής προστασία. Καμιά φορά οι ΙΠΑ βεβαίω αναφέρουν συγκεκριμένα κράτη-μέλη της Ένωσης και είχα υποβάλει γραπτή ερώτηση με έναν συνάδελφο που υποθέτω πως απάντησε η γενική σας διεύθυνση και η απάντηση είναι αηδίες αυτοί που μου στείλανε. Λέει πω η Κομισιόν προσπάθησε να διορθώσει τη λίστα το 1999 και το πάνελ του ΠΟΕ τότε είπε κάτι μπλα μπλα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί οι κυρώσεις να περνάνε ε, από το πάνελ του ΠΟΕ όμως είναι ένα πολύ σημαντικό διπλωματικό μέσο για τον εκπρόσωπο των ΗΠΑ για να ασκήσει πίεση σε μεμονωμένα κράτη-μέλη, για να σπάσει το σύστημα copyright της εσωτερικής αγοράς, που είναι ήδη κατακαιρματισμένο. Η βάση λοιπόν για τη δράση της Κομισιόν το 1999 ήταν πως δεν έχουμε εναρμονισμένη συμφωνία εφαρμογής εντός της Ένωσης και τώρα μου λέει η γενική σας διεύθυνση πως το 2004 έχουμε αρμονισμένα αστικά μέτρα οπότε κανένα πρόβλημα. Αλλά η ακόμα αναφέρουν τέσσερις χώρες κράτη-μέλη της Ένωσης ε, στην, έκδοση, στην έκθεση αυτή που έχουν ήδη εφαρμόσει την οδηγία του 2004 για τα πνευματικά δικαιώματα. Και είναι γνωστό πως η Ισπανία που επίσης ε, εφαρμόζει την οδηγία ξακολουθούσε να είναι στον κατάλογο το 2011 και έπρεπε να προχωρήσει πέρα από τα μέτρα της Ένωσης για να την αφαιρέσουν από τον κατάλογο. Και νομίζω πως επιγόντως η Κομισιόν πρέπει να χαράξει μια στρατηγική για να δει το τι θα κάνει με τις εκθέσεις αυτές. Αλλιώς δεν θα έχουμε μόνο εξαιρέσεις κατακαιρματισμένες αλλά και ένα κατακαιρματισμένο καθώς επιβολής. Και αυτό κατά την άποψή μου θα είναι μια κακή αρχή για την εποχή ε, την ψηφιακή. Οπότε σκοπεύετε να θέσετε αυτό το ζήτημα στη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Ε, ναι, είμαι ο τελευταίος ομιλητής. Εγώ. Έχω ε, δύο ερωτήσεις για τα θέματα για τις ε, σχέσεις εμπορικές με τις ΕΠΑ. Εγώ είμαι συντάκτης μαζί με έναν συνάδελφο μια επιστολής ε, που απευθύνθηκε σε Συμβούλιο και Κομισιόν και ενθαρρύνει την Κομισιόν να δει την πιθανότητα μιας φιλόδοξης συνθήκης με τις ΕΠΑ. Όμως στο γράμμα αυτό τονίσαμε την σημασία του να σεβόμαστε τα συγκεκριμένα συμφέροντα και ευαισθησίες της Ένωσης. Ήδη έχουν αναφερθεί γεωγραφικές ενδείξεις ε, τροφίμων, ε, επίσης προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ε, περιβαλλοντικές για τα φορτηγά κτλ. Τι ε, κάνει την Κομισιόν να πιστεύει πως οι ΙΠΑ οι οποίες πάντα ήταν πολύ αντίθετες ε, για λόγους αρχής με τα ζητήματα αυτά θα μπορέσουν στο τέλος να υποχωρήσουν. Και πώς θα μπορέσουμε να αποσπάσουμε υποχωρήσεις από τις είπα για τόσο ευαίσθητα ζητήματα. Χρειαζόμαστε νομίζω μία απάντηση. Νωρί. στο ζήτημα αυτό. Δεύτερη ερώτηση για την πολυμερή συμφωνία. Μας είπατε πως η Κομισιόν συμμετέχει στις αρχικές αυτές διαπραγματεύσεις και με το Συμβούλιο για την για τις συμφωνίες ε, ελευθεροπορίου. Πότε θεωρείτε πως θα, θα χρειαστείτε εντολή ε, διαπραγματευτική από το Συμβουλίο όταν θα έχετε τελειώσει τη διαπραγμάτευση ή κάπως νωρίτερα για να δει και την εντολή και το Συμβούλιο και να πει και κάτι και το Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, θα απαντήσετε σε αυτές. Α, δεν λοιπόν, θέλω να... Δεν θέλω να σας περιορίσω σε σχέση με, το, με τα ερωτήματα που θέλετε να θέσετε. Το ερώτημα του Ντανιέλ Κανσπάρη για την ένταση μεταξύ του διμερούς και του πολυμερούς τρόπου διαπραγματεύσεων. Και αυτό αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις βουλευτών. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε σχέση με πολυμερή διαπραγμάτευση μια συμφωνίας για τις υπηρεσίες. Αυτό ήταν και ένα από τα αιτήματά μας εξάλλου. Ήδη στη Γενέβη και στο Χονγκ Κονγκ. Εμείς είχαμε τονίσει ότι θα πρέπει να υπάρξει και κάποια μεγαλύτερη πρόοδος για τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις που να περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε μονάχα στα θέματα της γεωργίας και τέτοια θέματα. Δυστυχώς όμως, η μόνη διαβεβαίωση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι πρέπει για να γίνει αυτό μια πραγματικότητα πρέπει να έχετε και κάποιο συνομιλητή ο οποίο είναι έτοιμο να μιλήσει μαζί σα. Αλλιώ είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση χωρί συνομιλητή. Οι 20 αυτές χώρες που προανέφερα είναι έτοιμε να διαπραγματευτούν. Οι υπόλοιπε χώρες στα πλαίσια του ΠΟΕ δεν είναι έτοιμε. Ορθώς ή λανθασμένα, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι προφανώς εμείς θέλουμε αυτές οι διαπραγματεύσεις να ακολουθήσουν τους κανόνες του ΓΚΑΤ ώστε μετά να γίνουν, να μπορέσουν να πάρουν πολυμερή χαρακτήρα. Είναι διαφορετική η δομή από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ακολουθούν διαφορετική κατεύθυνση και δομή σε σχέση με τις διαπραγματεύσει συμφωνίες των υπηρεσιών, διαφορετική από αυτή τη δομή του ΓΚΑΤ, οπότε ακόμα και αν υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, πολύ δύσκολο να ενταχθεί μέσα σε ένα πολυμερές πλαίσιο θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή για μας, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε μέσα στην αρχιτεκτονική του ΓΚΑΤ. Το επιχείρημα των ΗΠΑ και άλλων χωρών θα μπορούσε να είναι ότι δεν είναι απαραίτητο σε ουσιαστικό επίπεδο να επηρεάζουν οι μορφές της συμφωνίας το, την ουσία. Αλλά με το να δουλεύει κανείς σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει γίνει δεκτό σε πολυμερές επίπεδο, έχει κανείς τη μεγαλύτερη δυνατότητα να προχωρήσει περισσότερο. Μπορεί να κρατήσει και να ξαναχρησιμοποιήσει κανόνες που να είναι είτε θετικοί ή αρνητικοί και να τους εφαρμόσει σε άλλα επίπεδα. Αλλά η διαδικασία του ΚΑΤ είναι αυτή η οποία προσωμιάζει περισσότερο και είναι πιο κοντά στην πολυμερή αντιμετώπιση. Κύριε Λάγκε, μου άρεσε η εικόνα αυτή που παρουσιάσατε για τα φορτηγά. Εμένα μ' άρεσαν πάντα την έβρισκα με τα αμερικάνικα καμιόνια. Είναι πολύ πιο ωραία από τα ευρωπαϊκά καμιόνια. Είναι τμήμα, αν θέλετε, του αμερικανικού ονείρου και του αμερικανικού πολιτισμού. και υπάρχουν απεικονίσει του ιδιαίτερα επιτυχή όχι μόνο από Αμερικανου αλλά και από Ευρωπαίου ζωγράφου. Αλλά η απάντηση στο δικό σα ερώτημα είναι η εξή. Θα μπορούν να εισαχθούν τα αμερικάνικα καμιόνια σε ευρωπαϊκές χώρες αν ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφέ, Αυτό είναι απλή ερώτηση. Αν αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να το δούμε. Αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα στον τομέα αυτό. Η κυρία Σάκε την έκανε, τουλάχιστον δεν είναι στην αίθουσα αυτή τη στιγμή, για την πρωτυποποίηση μια, ακολουθούμε μια διτή προσέγγιση από τη μία πλευρά. Ζητούμε από τους βιομηχανικούς κλάδους να παρουσιάσουν προτάσεις για το πώς θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδο στο δικό τους τομέα και αυτό είναι το τμήμα των διαδικασιών διαβούλευση που ξεκινάμε τώρα όλοι μαζί. Το, το κάνουμε αυτό γιατί νομίζουμε ότι είναι η προσέγγιση η οποία σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο είναι η πιο υποφελής και η πιο καρποφόρα, αλλά θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουμε και μια δομική προσέγγιση για το μέλλον. Να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο και είχαμε κάποιες επιτυχίες στο παρελθόν. Αλλά αυτό είναι μια χρονοβόρος και μακρά διαδικασία. Ενδιάμεσα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια κοινή δομή η οποία θα προωθήσει την προτυπωποίηση και για τα δύο μπλοκ συγχρόνως μια κοινή δομή. Πώς ακριβώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας το αναφέρω με λεπτομεριακό τρόπο αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε περισσότερη σκέψη για όλα αυτά, αλλά πρέπει να έχουμε κοινά εργαλεία για να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό. και μετά μπορείτε να σκεφτείτε ποιος μπορεί να είναι ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών για τέτοιες προσπάθειες τυποποίησης και προτυποποίησης και για τους κανονισμούς ακόμα θα μπορούσατε να ρωτήσετε τους εαυτούς σας κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει ένα δικαστικό σώμα που θα επιλύει τις διαφορές και το οποίο, στον οποίο μπορούν να προσφέρουν εταιρείες και Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα καιροτόμα και νομίζω ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερο καιρό για να μπορέσουμε να τα θεσπίσουμε αυτά και να τα υλοποιήσουμε και να τα βάλουμε στο κατάλληλο πλαίσιο. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι σε αμοιβαία βάση θα πρέπει να αποδεχθούμε τα πρότυπα και τους κανονισμούς επί τη βάση της αρχής με την οποία λειτουργεί η εσωτερική αγορά, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργήσει. Νομίζω ότι μια τέτοια πρόταση δεν είναι ρεαλιστική, δεν είναι εφικτή. για τις επιπτώσεις τώρα σε τρίτες χώρες. Υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την προσπάθεια αυτή. Ο κόσμος πράγματι αλλάζει, αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα και αν πράγματι θέλουμε να κρατήσουμε τη θέση μας, θα πρέπει να ενισχύσουμε ακριβώς τα επιχειρήματά μας. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, σεβόμενοι βέβαια τα ειδικά χαρακτηριστικά και των δύο ομάδων χωρών. Για τον κύριο Σαντό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να είναι μια σφαιρική συμφωνία. Αυτό που λέμε στα αγγλικά single undertaking. Και στα πλαίσια των συζητήσεων Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Πάντως η βασική ιδέα νομίζω ότι γίνεται δεκτή. Και νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός τρόπος να καταλήξουμε κάπου. Το να συμφωνήσουμε τώρα στους, δεσμούς, στους δασμούς και να αφήσουμε όλα τα άλλα στην άκρη ε, δεν είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Είναι πολύ περιορισμένα τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται δασμοί. Και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των συναλλαγών, στην ουσία καταλήγουμε σε πάρα πολύ υψηλά ποσά, γιατί έχουμε να κάνουμε με εκατομμύρια συναλλαγών και αν το κάνουμε αυτό τότε στην ουσία και από τις δύο πλευρές αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να επιδοτήσουμε τις βιομηχανίες μας και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να υπάρξει μια συνολικότερη συμφωνία έτσι ώστε η συμφωνία αυτή να μπορεί πράγματι να είναι λειτουργική. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Ζαντό ότι τα μη δασμολογικά τέλη δεν είναι τεχνικού τύπου, είναι μια πολιτική πραγματικότητα. Και υπάρχουν αρκετά θέματα στην Ευρώπη τα οποία αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα θέματα αυτά είναι τεχνικός. Παρόλα αυτά όμως η πραγματικότητα είναι πολιτική και δεν θα υπάρξει μεγάλη ευκολία για την εξέβρεση λύσης. Το αν αυτό θα επηρεάσει τον πολυμερή χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων. Προσωπικά εγώ είμαι υπέρ μιας πολυμερού συμφωνίας. D'essayer euh, de conclure des accords bilatéraux, c'est effort vraiment considérable. Οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτή τη φάση. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει συμφωνία για να προχωρήσουμε σε μια δεν υπάρχει συνένεση μάλλον για να προχωρήσουμε σε μια πολυμερή συμφωνία. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να προχωρήσει σε αυτή τη φάση. Το κρίνω εγώ αυτό, το κατακρίνω αν θέλετε. Θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά το λάθος δεν προέρχεται από τη δική μας πλευρά. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανοίξουμε κάποιες επιπλέον αγορές για τους παραγωγούς μας και για τις υπηρεσίες μας. Για τον κύριο Στέρντι, θέλετε να βάλουμε στην άκρη τη γεωργία, τον τομέα το γεωργικό. Έχετε πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Προτείνω να σας διορίσουμε πρέσβη εκεί για να τους πείσετε για την άποψή σας. Και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχετε πάρα πολλά και θετικά αποτελέσματα. για τις επιπτώσεις των εκλογών. Εγώ δεν θα ήθελα να εκφραστώ για τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Νομίζω ότι ο καθένας από όλους αυτήν την αίθουσα μπορεί να έχει τις δικές του προβλέψεις και το τι πιστεύω εγώ για τις εκλογές δεν θα προσφέρει κάθε, ε, κάποια προστιθέμενα αξία. Για τα TPP, Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εν μέρη πολιτικά εμπνευσμένο. Αυτό συμβαίνει με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου συχνά. Σχετικά με το TPP λοιπόν, η πολιτική συμφωνία προσδίδει μια, ένα μεγαλύτερο βάρος και δεν βασίζεται στην ίδια ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα σαν παράδειγμα των μεγάλων εμπλεκομένων στην ε, παγκόσμια οικονομία και των μεγάλων πρωταγωνιστών της γεωπολιτικής. Και γι' αυτό και η δική τους αντίληψη δεν είναι ταυτόσιμη με τη δική μας. Και εμείς προχωρούμε με τις χώρες του ΑΣΕΑΝ σε διαπραγματεύσεις και προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και με την Ινδία, να ξεκινήσουν οι επενδύσεις, οι συζητήσεις για τις επενδύσεις με την Κίνα, Όλα αυτά βασίζονται σε μία ανάλυση της κατάστασης καθαρά πολιτική. Το μέλλον θα δείξει ποια είναι η σωστή ανάλυση. Πάντως υπάρχουν πολιτικά θεμέλια στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Αλλά μία σωστή ανάλυση δεν μπορεί υποχρεωτικά να βασίζεται αποκλειστικά σε μία πολιτική ανάγνωση της κατάστασης. Θα δούμε, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα για τον κύριο Σόλτς. Υπάρχουν κάποιες διαφορές απόψεων οι οποίες σάπτονται της πίστης ή της μη πίστης στο ελόφερο εμπόριο. Δεν νομίζω ότι θα πείσω τον κύριο Σούλτς για την θέση μου. Τώρα δεν είναι εδώ έτσι κι αλλιώς, θα ήταν δύσκολο να τον πείσω. Αλλά ακόμα και αύριο ή του χρόνου αν τον συναντήσω, πάλι νομίζω ότι θα έχουμε μια διαφορά απόψεων η οποία να βασίζεται θα έλεγα σε θέματα αρχής. Νομίζω ότι η αποφυγή επικαλύψεων πράγματι μπορεί να μειώσει την απώλεια θέσεων εργασίας και σίγουρα εδώ ο ρόλος της οικονομίας κατ' εμέ είναι πολύ σημαντικός. Αλλά θα σταματήσω εδώ, στα πλαίσια της δημοκρατίας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Για τη συμφωνία λοιπόν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένε Πολιτείες παραπέμπω στη δήλωση του Βερολίνου για το κύριο Ντεζίρ για τα τέλη Αναφερθήκατε στη συμφωνία ναύτα, αλενά είπε ο κ. Ε, κάτι τέτοιο δεν μας επηρεάζει αυτή η συμφωνία, γιατί σε κάθε συμφωνία υπάρχουν ε, ξεχωριστοί κανόνες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο έτσι ώστε αυτοί οι κανόνες ελέγχου της προμήθειας, της προέλευσης συγγνώμη, των προϊόντων να μην επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένα σημαντικό θέμα και το οποίο θα πρέπει να ε, σεβαστούμε. Το ίδιο θα κάνουμε και στη συμφωνία με τον Καναδά. Ε, υπάρχει η δυνατότητα αυτή, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. για τις διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, όπου θέσατε αυτό το ερώτημα, αυτό το οποίο προβλέπετε είναι να εξαλειφθεί ένας αριθμός από να υπάρξουν κάποιες επιφυλάξεις ιδιαίτερα για τον οπτικο-ακουστικό τομέα και η βασική ιδέα του να ιδιωτικοποιηθούν ε, υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, αυτά δεν περιλαμβάνονται στους κανόνες του ΓΑΤ και επομένως για μας, για τους Ευρωπαίους θα διατυπώσουμε τις απαραίτητες επιφυλάξεις και έχουμε φυσικά την δυνατότητα να το κάνουμε και εγώ έχω καταγράψει τις ε, δεσμεύσεις οι οποίες έχουν γίνει Δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί είχατε αναφερθεί κύριε Ντεζίρ. Δεν μπορώ να σας δώσω αμέσως απάντηση. Μπορεί κανείς να έχει μία επιφύλαξη και να επιφυλαχθεί τη τελική του θέση μέχρι την τελική συμφωνία. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Κυρία Τεσσότερε, προσπαθήσαμε να βρούμε την απάντηση στο πάρα πολύ λεπτομεριακό ερώτημά σας. κατανοώ το ότι είσαστε προσιλωμένοι σε μια πιο στεναρή εφαρμογή της, ε, των κανόνων για την πνευματική ιδιοκτησία στο ίντερνετ παρά την αντίθεσή σας στο ΑΚΤΑ. Εμείς είμαστε κατά της ε, απαρίθμησης από τις ΗΠΑ κρατών μελών όπως η ΑΚΤΑ που συνάδουν με τις διεθνείς ε, Συμφωνίε για την πνευματική, για την πνευματική ιδιοκτησία, εφόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αντιμετωπίζουν με μονομένα τα κράτη μα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα περισσότερα. Συνεχίζουμε όμω συζητήσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε και εμεί έχουμε την, ε, Ηνωμένε Πολιτείε στη δική μα έρευνα για διάφορες με άλλες χώρες, όπως παραδείγματος χάρη για την Ιρλανδική μουσική, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να παράγουν εκθέσεις. Και για το τελευταίο ερώτημα του κύριου Μουρέιρα, όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, κύριε Μουρέιρα, εμείς λειτουργούμε από τη βάση της υφιστάμενης εντολής. Μπορεί εσείς να πιστεύετε ότι δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω εντολή. Αλλά φυσικά, εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι θα, υπάρξει, θα πρέπει να υπάρξει ένα ψήφισμα ή μια έκθεση ή οτιδήποτε ή και κάποια συγκεκριμένη εντολή. Βεβαίω μπορείτε να το πράξετε. Και θα πάρουμε τις παρατηρήσεις σας στα σοβαρά. Ξεκινάμε όμως από την θέση η οποία δεν διαφυσβητείται αυτή τη στιγμή από το Συμβούλιο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαπραγματεύση αυτής επί τη βάση της υφιστάμενης εντολή. Ξέρω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι προτού υπάρξει απόφαση για μια εντολή, θα πρέπει να δώσει και την θέση του, την γνώμη του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πρόκειται σε εσά να το κάνετε. Αλλά ίσως θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν με διαφορετικό τρόπο εφόσον πρόκειται για μια ήδη υφιστάμενη εντολή είτε με μια έκθεση, είτε με ένα ψήφισμα, όπως θέλετε να εκφράσετε τη θέση σας σε αυτήν την περίπτωση, αυτό είναι στη δική σα διακριτική ευχαίρεια, αλλά θα το χαιρετήσω κιόλα. θα το αποδεχθώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Ήταν πολύ παραγωγική η ανταλλαγή αυτή των απόψεων. Οπωσδήποτε θα επανέλθουμε στο θέμα. Ε, το αργότερο όταν θα συζητήσουμε την ε, έκθεσή μας με το ίδιο θέμα. Να αποχαιρετήσω τον κύριο Επίτροπο. Και ο χρόνος πιέζει, περνάμε στα θέματα 16 και 18. Θα γίνει μια κοινή συζήτηση για τρία σχέδια νομοδότησης. με στόχο τις λεγόμενες δημόσιες προμήθειες. για τις οποίες η κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή είναι η ΙΜΚΟ, αλλά μια που υπάρχει μια εξωτερική διάσταση ε, θα εκφέρει άποψη και η Επιτροπή μας. Η και για τις τρεις αυτές είναι ο Τζαν Λούκα σωστά από τους Σοσιαλδημοκράτε. στον οποίο δίνω και το λόγο. Τζαν Λούκα. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ιδιαιτέρως περιορισμένος. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Ξεκινώντας θα ήθελα να θέσω τα τυπικά, το χρονοδιάγραμμα κτλ. Υπενθυμίζω ότι η προστασμία για την κατάθεση της οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες είναι 18 Ιουλίου. Το να ζητήσουμε λοιπόν να γίνει μετακίνηση της συζήτησης για τις εκχωρήσεις το μήνα Σεπτέμβριο είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας καθυστερήσει. Η ψηφοφορία στην ίνκο βέβαια θα γίνει το Δεκέμβριο και έτσι θα μπορούσαμε και με την οδηγία για τις αναθέσεις και για τις δημόσιες συμβάσεις. Η έκθεση επί της ουσίας της ΣΥΝΚΟ έχει αλλοιωθεί θα έλεγα μέσω των τροπολογιών που ο ίδιος παρουσίασε. Καλό θα ήταν λοιπόν η γνωμοδότησή μας για την οδηγία για την ανάθεση συμβάσεων να μετακινηθεί έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία. Δεν θα επαναλάβω τώρα επί τη ουσίας αυτά τα οποία είχαμε πει στα πλαίσια μιας πρώτης παρουσίασης για το θέμα αυτό. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι μια ιδιαίτερα ανοιχτή αγορά, μια ανοιχτή αγορά κατά το 85% θα έλεγα, προς τρίτες χώρες. Παρ' όλα αυτά ζούμε σε έναν κόσμο στα πλαίσια του οποίου η πολιτική που ακολουθείτε δεν είναι να ανοίγουν οι αγορές στις δημόσιες συμβάσεις, η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις Ηνωμένε Πολιτείες, σαν παράδειγμα, είναι 12%, στην Ιαπωνία 23%, στον Καναδά 32% και 50% στην Νότια Κορέα. Ελπίζουμε ότι με την συμφωνία που υπογράψαμε ελευθέρων συναλλαγών θα βελτιωθεί η κατάσταση. Όλες αυτές λοιπόν χώρες έχουν ένα επίπεδο πρόσβασης γύρω στο 80-85%. Κινούμεθα λοιπόν προς μια κατεύθυνση η οποία να ορίζεται από τον ΠΟΕ, η οποία ρύθμιση ξεκίνησε ήδη από το 1981 συμμετέχει το σύνολο φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι και το πλαίσιο για την ρύθμιση των διεθνών αγορών στα πλαίσια της σύναψης δημόσιων συμβάσεων που αντιπροσωπεύουν το 3% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, αλλά μόνο για τις εμπλεκόμενες χώρες, οι οποίες είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση 32 χώρες και κάποιες περιφερειακές οργανώσεις χωρών. 27 είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βέβαια και παρατηρητές, δεν υπάρχουν άλλες, ε, είναι εκβιομηχανισμένες χώρες αυτές που συμμετέχουν, δεν υπάρχουν αναδυόμενες οικονομικά χώρες. Οι διαπραγματεύσεις βέβαια για την Κίνα είναι εν εξελίξη, το ίδιο και με την Ιορδανία και την Ουκρανία. Οι επιφυλάξεις τις οποίες έχουν θέσει οι μεγάλοι εμπορικοί εταίροι βέβαια έχουν το δικό τους βάρος. Έρχομαι τώρα στα συγκεκριμένα θέματα που θέτουν οι τροπολογίες που έχω εγώ καταθέσει και στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις και στην οδηγία των συμβάσεων των μεγάλων επιχειρήσεων νερού, ενέργειας, μεταφορών κτλ. Νομίζω ότι ιδιαίτερα η τελευταία οδηγία για την ενέργεια, τις μεταφορές, ε, τα ύδατα και η οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και παγκόσμιο βάρος. Έχουμε ζητήσει να υπάρχει μεγαλύτερη αμοιβαιότητα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων στα πλαίσια των διεθνών συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ φιλόδοξη για το άνοιγμα των διεθνών αγορών και γι' αυτό εμείς επιβεβαιώνουμε την αρχή της αμοιβαιότητας. Εδώ έχουμε αποδεχθεί την πρόταση Μπαρνιέ de Gucht προσαρμόζοντάς την στην τυπολογία της οδηγίας ε, την οποία έχουμε μπροστά μας. Δεν μιλάμε για κανονισμό αλλά για οδηγία, είναι κάτι το πιο γενικό λόγο. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να επιμείνουμε ε, στις ε, δημόσιες συμβάσεις που δεν καλύπτονται από διεθνείς συμφωνίες. Ακριβώς επειδή έχει προχωρήσει ο κανονισμός Barnier de στην οδηγία για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στα ύδατα, στην ενέργεια κτλ. και στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνονται αυτά τα οποία προϋπήρχαν στην προηγούμενη οδηγία ενισχύ για τις δραστηριοποιήσεις στον τομέα του ύδατος, ενέργειας κτλ. σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης των τρίτων χωρών αν οι οδηγίες πέρναγαν έτσι όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν πέρναγε ο κανονισμός Μπαρνιέ Ντεγκούχτ στην επόμενη σειρά, στον επόμενο γύρο νομοθετικών προτάσεων, τότε θα ήμασταν απολύτως ακάλυπτοι και γι' αυτό ακριβώς κατέθεσα μία τροπολογία η οποία επαναθέτει την αρχή της αμοιβαιότητας και η οποία εν πολλής επανέρχεται ε, σε αυτά τα οποία υπήρχαν στην προηγούμενη οδηγία για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς. Και επίσης ε, και η δυνατότητα για άμεσες εξαιρέσεις αν ε, το κόστος μιας πρότασης είναι χαμηλότερο κατά 50% από τις υπόλοιπες προτάσεις προσφορές όταν υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, ε, οι συγκεκριμένες μεγάλες διαφορές. Κάθε φορά που υπάρχει υποψία για υπερβολικά και ύποπτα χαμηλές προσφορές. Υπάρχουν συγκεκριμένα επίπεδα διεθνών ρυθμίσεων και σε σχέση με τη Σύμβαση 84 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τους κανόνες οι οποίοι θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί από πλευράς των οικονομικών εταίρων. Εμείς έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία εδώ με τους ε, συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι ασχολούνται ιδιαίτερα με τα θέματα της απασχόλησης, με τις κοινωνικές ρήτρε. Υπάρχουν και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται και με τις περιβαλλοντικές ρήτρε. Αλλά παρόλα αυτά η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να είναι προσεκτική στα σχέσεις στις εμπορικές με τρίτες χώρες και αυτές τις προηγούμενες αρχές τις οποίες προανέφερα τις κάνουμε δεκτές έγιναν δεκτές κατά 90 με 100% οι προτάσεις μου για τις λεγόμενες εσωτερικές διαδικασίες, in-house διαδικασίες. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα χρήσης ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων ε, για τις νέες ε, θεσμικές διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις εμπορικές ρυθμίσεις στα πλαίσια του Omnibus 1 και 2. Έχουν υπάρξει και αντιπαραθέσεις ε, με άλλες ε, συζητήσεις, μάλλον με άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έγιναν συζητήσεις, θα γίνουν και στο μέλλον συζητήσεις, ιδιαίτερα στα πλαίσια της οδηγίας για την καθυστέρηση των πληρωμών και για τις γενικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και από εμάς και στα πλαίσια επίσης ε, των ε, δημόσιων συμβάσεων σε σχέση με τον σεβασμό των ε, αποδεκτών συνθήκων εργασίας, των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Υπήρξε επίσης αναφορά στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει έτσι και λιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα λεγόμενα περιβαλλοντικά δικαιώματα, τα εργατικά δικαιώματα και στην εξαίρεση του κριτηρίου του χαμηλούμενου κόστους. Εδώ είναι κάτι το οποίο απασχολεί τον εισηγητή της ΣΥΝΚΟ, τον κύριο Ταραμπέλα. Σαν να μην είναι το μοναδικό κριτήριο επί τη βάση του οποίου λαμβάνεται η απόφαση για την σύναψη δημόσιας σύμβασης. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους κύριους εισηγητές από το ΑΕΛ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα μιλήσω εξ ονόματος της κυρίας Χάνσλικ, η οποία είναι η σκιώδης εισηγήτρια και θα μιλήσω πολωνικά. Sorry. E, pani Hanzik, pragnie podziękować panu słusznie za propozycję. Ευχαριστώ. Κυρία Χάνσλικ, θα ήθελα να τον κύριο Σούστα για το σχέδιο έκθεσης ε, και τις ε, τροπολογίες γιατί θεωρεί πως πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζει να μην ε, έχουμε προβλήματα στη συμβεσμούς αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελε να τονίσει πρώτα απ' όλα συνδέονται με τους όρους ε, των ε, ΣΔΙΤ συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα γιατί ο τρόπος ε, με τον οποίο έχουν συνταχθεί από την Κομισιόν δεν δίνει την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την εξαίρεση γιατί υπάρχει υψηλότερο ποσοστό δραστηριοτήτων που προτείνεται οπότε θα προτιμούσε η διάταξη αυτή να διατυπωθεί με έναν τρόπο που θα ικανοποιεί την απόφαση του ΔΕΚ γιατί το ΔΕΚ μιλάει για ουσιαστικό τμήμα των δραστηριοτήτων και δεν πρέπει να πάμε παραπέρα από αυτά τα οποία λέει το δικαστήριο και δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε το εάν, να δούμε το εάν το ουσιαστικό κομμάτι είναι 89% ή 90% όταν μιλάμε δε για την αρχή της αμοιβαιότητας πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί γιατί η ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων προμηθειών παραμένει πιο ανοιχτή σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει να διασφαλίσουμε και ένα σημαντικό μερίδιο για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως να μην υπάρχει διακριτική μεταχείρισή τους και να τονίσουμε το ότι πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία και να δρούμε τρόπο προσεκτικό. Σκοπεύουμε λοιπόν να εξαιρέσουμε, η πρότασή μας είναι να εξαιρεθεί η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 4. Δημόσιε προμήθειε για κοινωνικέ υπηρεσίε γιατί η κυρία Χάντσλεκ βεβαίω γνωρίζει πως έχουμε διαφορετικό κανονισμό στον τίτλο 3 αλλά φαίνεται πως κάτι τέτοιο είναι εκτός των ε, αρμοδιοτήτων μας. Η κυρία Χάνσλιτ λοιπόν θα ήθελε να παρουσιάσει κάποιες ε, τροπολογίες όταν μιλάμε για εξαιρετικά χαμηλές ε, προσφορές. Είναι σημαντικό να το δούμε αυτό και καλό είναι το ότι η Κομισιόν προτείνει κάποιες ειδικέ προβλέψεις. Θεωρούμε όμως πως η πρόταση της ε, Κομισιόν πρέπει να είναι πιο λεπτομερής. Γι' αυτό θα καταθέσει και σχετικές τροπολογίες η κυρία και Επίσης, οι υπερβολικά χαμηλές ε, τιμές είναι κάτι το οποίο αναφέρει ο εισηγητής, αλλά όταν μιλάμε για τουλάχιστον πέντε προσφορές δεν ξέρουμε αν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο οπότε θα προτιμούσε η κυρία Χάντσλικ να διαγραφεί ευχαριστώ η Ζαντό από τους Πράσινους ε, ο εισηγητής εδώ προτείνει να αναβάλουμε τη συζήτηση για τις δημόσιες προμήθειες γιατί όχι αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι εμεί πρέπει να βασιστούμε στην προηγούμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ανεκρίθη τον Οκτώβριο για το θέμα αυτό, που λέει σαφώ ότι δεν υπάρχει ανάγκη να ξεκινήσουμε νέα διαδικασία για τα θέματα αυτά, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν διακρίσεις και στρεβλώσεις <clears throat> σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ότι η μία αναθεώρηση της ε, οδηγίας δεν έχει νόημα όταν δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί και διακριβωθεί στρεβλώσεις οι οποίες θα μας υποχρεώνουν ακριβώς να προβούμε σε μια τέτοια τροποποίηση της οδηγίας. Επομένως, είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο που αποτελεί τη βάση μας. Θα πρέπει επί τη βάση αυτής της θέσης να αξιολογήσουμε την ανάγκη τροποποίησης της οδηγίας. Για τα άλλα θέματα τώρα, τα άλλα στοιχεία κατανοώ πολύ καλά την θέληση να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης αμοιβαιότητας. Και αυτό ανταποκρίνεται σε ένα θεμητό πολιτικό στόχο. Για μας όμως δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει τον πυρήνα των τροπολογιών που θα καταθέσουμε. Υπήρξε η συζήτηση προηγουμένως που αφορούσε την ε, διατλαντική σχέση η ισχύ των Αμερικανών στην εμπορική πολιτική τους είναι ότι η εμπορική τους πολιτική βασίζεται σε μια βιομηχανική πολιτική και σε μια αγροτική πολιτική που είναι σαφής και στεναρές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια αγροτική πολιτική και μπορεί αυτό να μην αρέσει στο Ρομπέρ, αλλά αυτές έχουν, αυτή η πολιτική έχει κάνον, έχει διαμορφώσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν έχουμε καμία βιομηχανική πολιτική. Επομένως, όταν μιλάμε για το εμπόριο, το ερώτημα είναι τι θέλουμε να υποστηρίξουμε, τι θέλουμε να προασπίσουμε. Νομίζουμε ότι η πολιτική μας για τις δημόσιες αγορές, επειδή αναφέρθηκε το θέμα αυτό, αυτό είναι μια πολιτική που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας μας. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο με την Νότια <clears throat> Κορέα ή τον Καναδά, αλλά μιλάμε για 18-19% της συνολικής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν στο τομέα αυτό, όταν μιλάμε για τις δημόσιες προμήθειες και αγορές, θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να έχουμε για τις οικονομίες μας και μετά να δούμε ποια είναι η σωστή υλοποίηση σε εμπορικό επίπεδο αυτής της πολιτικής. Εμείς ως οικολογοί, οικολογοί θεωρούμε ότι η προτεραιότητα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρόκειται μονάχα για την δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, αλλά και για τη δυνατότητα πρόσβασης και στις ευρωπαϊκές αγορές και προμήθειες. Το ίδιο ισχύει για την πτυχή του περιβάλλοντος. Οπότε αυτό είναι αντίθετο με αυτά τα οποία λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς τονίζουμε την ανάγκη του τοπικού περιεχομένου. Έχουμε μια σύγκρουση με τον Καναδά για το θέμα του Οντάριο στην Ιταλία υπάρχει μια πολιτική για τι ανανεώσιμε ενέργειε που βασίζεται στο τοπικό περιεχόμενο. Εμεί ω πράσινοι θεωρούμε ότι έχουμε ελάχιστα εργαλεία βιομηχανική πολιτική σήμερα, <clears throat> ελάχιστα εργαλεία τα οποία δεν θα ήταν πολυδάπανα και γι' αυτό η πολιτική για τις δημόσιες αγορές θα πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο της βιομηχανικής μας πολιτικής, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η έννοια του τοπικού περιεχομένου θα έπρεπε να είναι από του κύριου άξονες της βιομηχανικής μας πολιτικής στην Ευρώπη και επομένως και τους άξονες της εργασίας μας. Η κυρία Μακκλάρκιν έχει το λόγο από τους συντηρητικούς. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πάρα πολύ σημαντικό έργο και το δύσκολο έργο που οδήγησε σε, αυτές τις σε αυτή τη γνωμοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο ένα πλαίσιο για τι δημόσιε προμήθειε, ώστε να ανακλά καλύτερα τι ανάγκε που έχουμε σήμερα και με στόχο να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει να λάβει υπόψη το συνολικό πλαίσιο τη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε. <clears throat> θα ήθελα σχετικά να αναφέρω ορισμένα θέματα στον εισηγητή σε σχέση με τα κατόφλια για τι συμβάσει παραχώρηση Ξέρω ότι ο εισηγητής έχει προτείνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των αγαθών και των υπηρεσιών με όριο 2,5 εκατομμύρια για τις υπηρεσίες και 5 εκατομμύρια για τις άλλες συμβάσεις. Θα ήθελα να ξέρω γιατί ο εισηγητής προτείνει αυτή την διαφοροποίηση και αν βασίζεται στην ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να κάνει τις δημόσιες προμήθειες πιο πολύ δάπανε. Δεν ξέρω αν έχει κάποια συγκριτικά στοιχεία τα οποία ε, αναφέρουν τι επίπτωση θα έχει αυτή η αλλαγή των κατοφλίων και ίσως και η Κομισιόν έχει κάποια σχόλια για τις δυνητικές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών. Επίσης θέλω να ζητήσω τον εισηγητή για ορισμένε συγκεκριμένε τροπολογίες 4, 5 και 23 στον κανονισμό για τις δημόσιες συμβάσεις. Εκεί γίνεται μνήα στα εργαλεία αμοιβαιότητα της Κομισιόν Όλα αυτά δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα στο νομοθετικό πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν. Εδώ θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το να αναφέρουμε ρήτρε του ίδιου του κανονισμού για τι δημοσίε προμήθειε, γιατί μπορεί να επιφερθούν αλλαγέ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για μένα και έχουμε πολλά να πράξουμε από την πλευρά της Επιτροπής μας. Ελπίζω ότι ο εισηγητής θα μπορέσει να λάβει υπόψη όλες αυτές τις ανησυχίες μου. Σας ευχαριστώ κύριος Κασπάρη από το ΕΛΚ. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα ήμουν ευγνώμων ο εισηγητής μας να ξανασκεφτεί ορισμένες τροπολογίες. Επί της αρχής μπορώ να υποστηρίξω αυτά τα οποία γράφει και επί της ουσίας δεν έχουμε μεγάλες διαφορές. Αλλά δύο πράγματα θέλω. Το ένα είναι το θέμα αρχή, το ποιε είναι οι αρμοδιότητε μα ω Επιτροπής και δεύτερον το θέμα της εξωτερικής διάστασης των δημοσίων προμηθειών όπου υπάρχουν αρκετέ τροπολογίες και είναι ακριβώ ο τομέας όπου έχει την κύρια αρμοδιότητα η Επιτροπή μας και πραγματικά εγώ έχω πρόβλημα με την εξωτερική διάσταση στις τρεις αυτές εκθέσεις. Θα πρέπει νομίζω να συμφωνήσουμε σε μια λογική λύση γιατί θα συζητήσουμε και τη δική μου έκθεση αλλά μετά δεν έχουμε το βασικό ρόλο. Εμείς θα υποβάλουμε γνωμοδότηση στην ΙΜΚΟ η οποία θα κάνει ό,τι θέλει και κρίμα είναι μετά η ΙΜΚΟ να αποφασίσει κάτι για την εξωτερική διάσταση ε, το οποίο δεν θα ταιριάζει με τις δικές μας ιδέες που θα επεξεργαστούμε στη δική μου έκθεση. Γι' αυτό η παράκλησή μου να σκεφτεί ο εισηγητής και όλοι μας μήπως αυτός ο τομέας της εξωτερικής διάστασης όταν μιλάμε για κάποιες εξωτερικές εταιρείε να μπορέσουμε να τις αποκλείσουμε και να το βγάλουμε αυτό το κομμάτι εκτός στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κυρίων και να πάει στη δικιά μου την έκθεση. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, δεν θέλω να την αποφύγουμε και θα πρέπει να συμφωνήσουμε, αλλά σας παρακαλώ να συμφωνήσουμε εμείς εδώ πέρα και να μην το δώσουμε στην ΙΜΚΟ. Γιατί δεν είναι δική τους αρμοδιότητα. Παρακαλώ λοιπόν να γίνει αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο της δικής μου έκθεσης και πραγματικά θα ήμουν αν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Σωστό λέει ο πρόεδρος. Μπέρντ Λάγκε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Χωρίς αμφιβολία οι δημόσιες προμήθειες είναι στρατηγικός μοχλός για τη βιομηχανική πολιτική και έχουμε βεβαίω και την βιομηχανική πολιτική που πρέπει να συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο και θεωρώ πως πρέπει και εδώ να διατυπώσουμε αφενός το ότι ε, κατά κύρωση δημοσίων προμηθειών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές ανάγκες, δηλαδή τις περιβαλλοντικές ε, προδιαγραφές, δηλαδή φορτηγά και λεωφορεία να πληρούν τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να τονίσουμε το ζήτημα της καινοτομίας. Π.χ. τα PC που αγοράζουμε να προωθούν και το περιβάλλον. Οι ΕΠΑ, παραδείγματος χάρη, έχουν ορίσει ποσοστώσεις καινοτομίας στις δημόσιες προμήθειες. Οπότε θεωρώ πως πρέπει και εδώ πέρα να ε, γράψουμε σαφώς πως πρέπει να υπάρχει και ένα κριτήριο πολιτικής βιομηχανικής και βεβαίως και μια εξωτερική διάσταση. Ανεξαρτήτως την έκθεση την οποία θα παρουσιάσετε εσείς εδώ πέρα, γιατί αυτά είναι τα κριτήρια τα οποία ε, θα ισχύσουν συνολικά για τις δημόσιες προμήθειες και νομίζω πως οπωσδήποτε είναι και προς το συμφέρον της προστασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να έχουμε κάποια κριτήρια για εξωτερικές εταιρείες. Παραδείγματο χάρη το ζήτημα κοινωνικών, περιβαλλοντικών προδιαγραφών, το ζήτημα παράνομης επιδότησης και οπωσδήποτε και το θέμα της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν έχω καμία όρεξη να ε, αγοράζουμε προϊόντα τα οποία παραβιάζουν ε, την πνευματική διοκτησία από τρίτες χώρες. Αυτό πρέπει να μπουν στα κριτήρια. Νομίζω μπορούμε να το κάνουμε ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με τις δημόσιες προμήθειες από εταιρείε ε, τρίτες. Μάλιστα, ας ακούσουμε τώρα την Κομισιόν για να κλείσει αυτή η συζήτηση. Σύντομα, παρακαλώ, ποιος θα εκπροσωπήσει την Κομισιόν. Η κυρία Τζανέτη από την Γενική Διεύθυνση της Αγοράς. Και τα τρία θέματα μαζί. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Ένα θέμα θα ήθελα να υπογραμμίσω, το οποίο έχει ήδη τεθεί στη συζήτηση, το θέμα της αμοιβαιότητας. Ξέρετε ότι εμένουμε εμεί σαν Επιτροπή στην αμοιβαιότητα. Και γι' αυτό καταθέσαμε μία πρόταση για το μέσο, για τις δημόσιες, το διεθνές μέσο για τις δημόσιες προμήθειες. Νομίζω ότι αυτό έγινε μετά από συζητήσεις οι οποίες έγιναν. Είναι ε, αλήθεια ότι κατανοώ τις ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί για το χρονοδιάγραμμα ανάμεσα στις δύο προτάσεις, δηλαδή τις συμβάσεις παραχώρησης από τη μία και τις δημόσιες συμβάσεις από την, άλλο, από την άλλη, αλλά ανήκουν σε ένα συνολικότερο, ευρύτερο πακέτο. Πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν σωστό να επικαλύψουμε τις ρυθμίσεις και να εισάγουμε και να εξάγουμε προβλέψεις και ρήτρε από το ένα μέσο στο άλλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να γεφυρώσουμε το κενό χρόνο ανάμεσα στα δύο α, επιμέρους θέματα στα πλαίσια ενός πακέτου. Αυτό είναι σημαντικό για να μην αποστέλουμε και ε, μηνύματα συγχύσεως προς τους διεθνείς εταίρους μας. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα μεγαλύτερο πακέτο, προσωρινά κρατώντας το status quo, το ισχύον καθεστώς όπως υπάρχει, περιμένοντας να τεθούν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Θα μπορούσα να είμαι λεπτομερέστερη στα επιμέρους θυμία, αλλά νομίζω ότι ίσως τώρα πια δεν είναι η κατάλληλη στιγμή και ίσως να απαντήσω σε ερωτήσεις τις οποίες θα θέλατε να σας θέσω. Να μου θέσετε, συγγνώμη. Το θέμα των ανωτάτων ορίων. τα διάφορα όρια, οι διαφορές στα όρια στον τομέα των υπηρεσιών σαν παράδειγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες. Ξέρετε ότι η ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης είναι κάτι το ιδιαίτερος περίπλοκο. Είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί περαιτέρω και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και να ακολουθήσουν ορισμένες αλλαγές στις προτάσεις τις οποίες κάνουμε. Ο εισηγητής μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις στις παρατηρήσεις που έγιναν. Και στον κύριο Κάσπαρη. Κύριο Σέστα, ευχαριστώ. Εγώ στην εισαγωγή δεν αναφέρθηκα για λόγους χρόνου στο ιστορικό των συζητήσεων μέχρι τώρα. Για να είμαι σαφής, σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Κάσπερ υπάρχουν δύο εναλλακτικέ. Έχει δίκιο σε αυτό και εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρήσω ότι θίγομαι, ότι προσβάλλομαι. Αλλά η πρόταση Κάσμαρη είναι να μην προχωρήσουμε στη γνωμοδότηση. Αυτό θα μπορούσε να είναι σωστό από μία άποψη, αλλά από την άλλη θα πρέπει η Επιτροπή ίντε να το αποφασίσει αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Τα βασικά θέματα που περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση και οι βασικές τροπολογίες άπτονται έμεσα ή άμεσα των διεθνών συνεπειών αυτών των ρυθμίσεων. Να κάνω την αντίθετη εδώ επιχειρηματολογία. Ποιες είναι οι πλευρές μέσω των οποίων επιχειρήσεις τρίτων χωρών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αθέμητα μέσα ανταγωνισμού τα χρησιμοποιούν για να κερδίσουν προμήθειες. Ε, σαν παράδειγμα μη, σεβαστός, μη σεβασμός της ποιότητας, μη σεβασμός των, των προβλέψεων και των προτύπων ασφαλείας, μη σεβασμός των περιβαλλοντικών προβλέψεων, ε, πολύ ε, χαμηλές προσφορές και εκεί όπου υπάρχουν ε, υποψίες σε σχέση και με τα πλαίσια με τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε τα τοπικά συμφέροντα, γιατί όπως είπε ο Ζαντός σωστά δεν κοιτάμε μόνο τα εσωτερικά θέματα, αλλά κοιτάμε και τα εξωτερικά. Για τις προτάσεις της συγκεκριμένες Μπαρνιέντε Γκούχτο, για τις οποίες είναι εισηγητής ο κύριος Κάσπαρη. Πράγματι εκεί έχουμε μια άλλη ευκαιρία. Έχουμε μια άλλη δυνατότητα και θα πρέπει να σταθούμε ε, προσεκτικοί θα έχουμε μπροστά μας ένα νομοθετικό σενάριο το οποίο θα πάρει την εξή μορφή. Το λέω αυτό στον Κασπάρη γιατί θα συζητήσουμε και τον κανονισμό de Gucht Barnier. Οι δύο αυτές οδηγίες, δημόσιες συμβάσεις και οι δραστηριοποιούμενες στους τομείς ύδατος, ενέργειας κτλ. Συν πιθανώς την οδηγία για την ανάθεση παραχωρήσεων είναι οδηγίες οι οποίες θα γίνουν δεκτές θα γίνει δεκτός, το αν θα γίνει δεκτός ο κανονισμός Μπαρνιέ Γκούχτ έχω πολλές αμφιβολίες. Θα το συζητήσουμε, θα αντιπαρατεθούμε, θα, αλλά έχω αμφιβολίες για το αν θα καταλήξουμε. Εγώ δεν έχω καν καταλάβει ποια θα είναι η αρμόδια επί της ουσίας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και δεν έχω επίσης καταλάβει και ποια είναι η κοινή θέση των Μπαρνιέ Γκούχτ σε σχέση με τον κανονισμό αυτό. Το να είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι οι οδηγίες αυτές θα γίνουν δεκτές χωρίς να εντάξουμε στις οδηγίες αυτές την αρχή της αμοιβαιότητας, θα καταλήξουμε με οδηγίες ιδιαίτερα στις δραστηριοποιούμενες του τομείς του ύδατος ενέργειας και στις δημόσιες συμβάσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα τις εκθέσουμε σε τομείς ευαίσθητους όπως οι υπηρεσίες, όπως ε, όλες ε, θα έλεγα κοντινές στον πολίτη υπηρεσίες οι οποίες δεν καλύπτονται και δεν προστατεύονται από τον ανταγωνισμό των τρίτων χωρών. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί λοιπόν ή θα είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουμε στα πλαίσια μιας συνολικής νομοθετικής ρύθμισης και όχι μόνο Μπαρνιέ Γκούχτ ή δεν θα έχουμε κανένα σύστημα προστασίας, προστασίας όχι με την έννοια του προστατευτισμού αλλά ελέγχου. Λοιπόν, δύο επιμέρους απαντήσεις για τις υπηρεσίες. Η ποια είναι η διαφοροποίηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στις αναθέσεις παραχωρήσεων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, την κοινωνική βοήθεια και την υγεία. Είναι τομείς πάρα πολύ ευαίσθητοι. Δεύτερο, για τα λεχόμενα in-house 100%. Κοιτάξτε, αν κάτι γίνεται εσωτερικά, in-house, τότε είναι κάτι που γίνεται εσωτερικά. Ο λίγων εσωτερικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει. Και μια τελευταία απάντηση προς τον κύριο Ζαντό. Πιστεύω ότι η ανάγνωση των τροπολογιών τις οποίες θα καταφέσουν οι συνάδελφοι θα μου επιτρέψουν να καταλήξουμε σε μια καλύτερη μορφή συντονισμού μεταξύ μας. Υπενθυμίζω όμως τον κύριο Ζαντό ότι στο κείμενο των προτάσεων για τις οδηγίες ορισμένα από τα θέματα τα οποία τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα ε, σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανάτατα όρια, σε σχέση με τη δυνατότητα συνέχισης των διαπραγματεύσεων, περιλαμβάνονται στις οδηγίες και οι οδηγίες στην ουσία διευρύνουν τις δυνατότητες αυτές. Όπω και να έχουν τα πράγματα, ότι εγώ θα περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις τροπολογία και μαζί με τους συντονιστές θα μπορέσουμε να συντονιστούμε και να σεβαστούμε βέβαια τις βασικές αρχές που θεμελιώνουν το σύνολο αυτών των προτάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, θα πρέπει να το σεβαστούμε. Προθεσμοί για τις τροπολογίες, για τις δύο οδηγίες, για τις δημόσιες ε, ε, συμβάσεις και, και κοινοφελείς υπηρεσίες 18 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα και σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις παραχωρήσεις, παραχωρήσεις παραχωρήσεων θα την επανεξετάσουμε το Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει λοιπόν χρονοδιάγραμμα για τροπολογίες ακόμα. Πρώτο ήρθα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης να σας ε, θυμίσω ότι βάσει της απόφασης των συντοριστών η προθεσμία για τις τροπολογίες για, την, για το λεγόμενο πρωτόκολλο ΆΤΑ μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ είναι η 16 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. 16 και 6. 16 Ιουλίου, 6 το απόγευμα. Τελευταίο στοιχείο είναι δύο στοιχεία που θα τα αντιμετωπίσουμε από κοινού τα σημεία 19 και 20 για κανονισμούς που εισάγουν στην Ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποφάσεις της, ε, τους εναρμοσμένους κανόνες της ε, Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την ε, Ευρώπη σε σχέση με πρότυπα για αυτοκίνητα οχήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί βασιζόμαστε όλο και περισσότερο στα διεθνή πρότυπα για τα αυτοκίνητα οχήματα όπως έχουν καταρτιστεί από τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι ένα σημαντικό τρόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει πίεση στους εμπορικούς μας εταίρους. Αυτό κάνουμε με την Ιαπωνία και ελπίζω να το κάνουμε και με τις Ηνωμένε Πολιτείε με στόχο να τους πιέσουμε να υιοθετήσουν τα ίδια πρότυπα και με, σωστή, με ισχυρή επιχειρηματολογία γιατί έτσι δεν θα υιοθετούν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά διεθνή πρότυπα τα οποία θα είναι πλέον από κοινού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Εγώ είμαι και ο εισηγητής για τα δύο θέματα παρεπιπτόντω και έχω μια πολύ θετική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ στεναροί για τα θέματα αυτά. Το σημαντικό λοιπόν, το θέμα αυτό δεν είναι ένα θέμα ίσονος σημασίας, δεν έχω ακόμα χρονοδιάγραμμα. Προτείνω να έρθουμε για μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο. Έχουμε καιρό. Αλλά μην θεωρήσετε ότι αυτό είναι ένα θέμα περιθωριακό. Είναι σημαντικό γιατί αυτό ενισχύει την ικανότητά μας διαπραγματεύσεων με τους ισχυρούς εταίρους μας για την ισχυρή αυτοκινητοβιομηχανία, ιδίως της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλει κανείς να λάβει το λόγο. Όχι. Οπότε θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ποιος θα λάβει το λόγο από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Η Μαργαρίτα Τελρομάου Λοβρόζου. Ποιος θα μιλήσει. Ναι κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι εδώ. Εδώ είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ βεβαίως. Δεδομένης της ώρας θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Είναι θετικό ότι γίνεται η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή ήδη επί των δύο αυτών προτάσεων που όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος είναι πράγματι πολύ σημαντικές. στο διεθνές πλαίσιο. Και πράγματι, οι δύο αυτές προτάσεις υποβάλλονται τώρα λόγω αλλαγών στην συνθήκη από το 97 μέχρι σήμερα και το 2000 μέχρι σήμερα. Οπότε πρέπει να προσαρμοστούν και τα κείμενα αυτά στη συνθήκη. και στις διαδικασίες υιοθέτηση και σύναψης διεθνών συμφωνιών. Βεβαίω το κείμενο μιλάει ακόμα για σύμφωνη γνώμη, αυτά πρέπει να διορθωθούν. Και βεβαίω και τη θέση που πρέπει να υιοθετήσει η Ένωση σε ένα φορέα που έχει συσταθεί με βάση τη Διεθνή Συμφωνία. Το άρθρο 289 τώρα βεβαίω έχει μια απλούστερη διαδικασία που πρέπει να συμπεριληφθεί στα δύο κείμενα και κάποιες άλλες παράγωγες νομικές βάσεις. Και όλα αυτά θα διορθωθούν στο κείμενο. Το άρθρο 44 θα διαγραφεί και το κείμενο θα ευθυγραμμιστεί με τις συνθήκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό τον Οκτώβριο. Αυτά. Για σήμερα αποφάσισα να αναβάλω το σημείο 21 για αύριο. Αύριο λοιπόν. Αύριο δεν θα συνεδριάσουμε σε αυτή την αίθουσα. Στο ίδιο κτίριο, αλλά στον πέμπτο όροφο. Τα λέμε αύριο Γεια σας.